Dear colleague, please, we have to go. The agenda is very busy today, so please. Uh, Παρακαλώ να καθίσετε γιατί θα ξεκινήσουμε και έχουμε πολύ πλήρες πρόγραμμα σήμερα. Βλέπω ότι είσαστε όλοι έτοιμοι, άρα ξεκινάμε τις ψηφοφορίες η ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος που αφορά ε, στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην έκθεση για τη Μακεδονία το 2010 ο κύριος Τάλερ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ε, τροπολογίες υπαριθμών 11. Ο κύριος Κούκαν θέλει να παρέμβει. Θα σταματήσουμε να στείλουμε λιγάκι την ψηφοφορία για να παρέμβει ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ. Πριν να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ να θέσουμε σε ψηφοφορία μια προφορική τροπολογία που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι και που αφορά τη μνήμα του ονόματος Μακεδονία στο κείμενο του ψηφίσματος. Η πρόταση είναι να αλλάξει η ονομασία Μακεδονία εκεί που αναφέρεται στο κείμενο και να αναφέρεται το όνομα πρώην, δημοκρατική, πρώην, δημοκρατία της Μακεδονία, πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ΦΥΡΟΜ δηλαδή, και όλες οι αναφορές στη Μακεδονία θα πρέπει να αντικατασταθούν από το πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Καλώς, αν δεν υπάρχουν και συμφωνεί και ο εισηγητής, απέχει ο εισηγητής. Καλώς, ο κύριος Λάμστορφ. Δεν ξέρω τι ακριβώς προβλέπει το καταστατικό, κατά πόσον επιτρέπεται η προφορική τροπολογία ή κατά πόσον αρκεί ε, να διαφωνήσει ένας για να μην εγκρίνεται μια τροπολογία. Αν ισχύει το τελευταίο, εγώ διαφωνώ με αυτήν την ε, προφορική τροπολογία που μόλις ετέθη. Άρα δηλαδή ε, αρκεί ένας ε, να διαφωνήσει, δεν χρειάζεται να διαφωνήσει κι άλλοι. Εσείς διαφωνείτε, άρα ε, περνάμε στην επόμενη, τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, παρακαλώ ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την τροπολογία 11 άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν όλοι. Δέκα συνάδελφοι ακόμη δεν έχουν ψηφίσει. Παρακαλώ ψηφίστε. Βλέπω να έχουν μπει οι κάρτες, αλλά δεν βλέπω την ψηφοφορία, το αποτέλεσμα. Λήξη της ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 13 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 15 τροπολογία 15 Είναι συμβατή 14, 14. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Οπότε πηγαίνουμε στη δεύτερη συμβαστική τροπολογία σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Αβέβαια το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ για επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 28. Τέλος ψηφοφορίες. 24 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. Ποιο είναι υπέρ τη συμβαστική ε, τροπολογία 3 κατά αποχέ εγκρίνεται. 37 τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 42 υπέρ. Διορθώνω λέει ο πρόεδρος και την 40 πρέπει να ψηφίσουμε γιατί την 39 δεν εγκρίναμε. Ποιος είναι υπέρ, 40, 40 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 41, ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Σαράντα εννέα κάποιος ζήτησε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της 49. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 49. Τέλος ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. 51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ με την προφορική τροπολογία κούκαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 74 έχει αποσύρθει. 73 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ. Για το πρώτο κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 78 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 82 κατά ασαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την τροπολογία 82 άρχεται η ψηφοφορία Chiusa la votazione elettronica. Τέλος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 26 no, 23 sì. Απορρίπτεται 23 υπέρ, 26 κατά. 83. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 με την προφορική τροπολογία Κούκαν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ ηλεκτρονικό έλεγχο θέλετε για την 88 Πολύ ευχαρίστως. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 88. 88. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίες. 40 υπέρ, 11 κατά, μία αποχή. Έγκρινεται. 89. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 90. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96. Ποιος είναι υπέρ. Με διορθώνει η γραμματεία ότι πρέπει να ψηφίσουμε και την 94 και την 95. 94 πρώτα λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ της 94. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 και 98 είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Όχι, πλάκα κάνετε. 97-98 ποιος είναι υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Ah, είναι 99 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 τροπολογία υπέρ. Κατά. Μάλλον απορρίπτεται. Αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 110. 110 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 29 21 υπέρ, 33 κατά. Απορρίπτεται. 108. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 119, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 127, υπέρ, ή μάλλον 123 διορθώνει ο πρόεδρος. 123 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 136 με προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Γι' αυτό ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 137. Τέλος. 29 κατά 25 υπέρ. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές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 αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή μάλλον εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρο. Αιτιολογική σκέψη α. Τροπολογία 2. ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ, Μάλλον εγκρίνεται. Τροπολογία 3. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η κυρία Γιαννάκου. Ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία 5 θα μπορούσα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία. Είναι στη δική μου τροπολογία η προφορική. Θα πρότεινα να διαγράψουμε ιδιαίτερα της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων μάλλον. Ιδιαίτερα των κυβερνήσεων. Especially of the governments. Αυτό μπορούμε να το διαγράψουμε το ιδιαίτερο των κυβερνήσεων, especially of the governments. Και λέει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και των, των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των κοινοτικών κρατών, κοινοτικών κρατών μελών. Αυτή είναι η πρότασή σα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει για την προφορική τροπολογία μπορούμε να την ψηφίσουμε. Υπάρχει όμω μια αντίρρηση από ό,τι βλέπω ή όχι. Όχι, όχι, δεν είναι αντίρρηση, δεν είναι έσταση. Δεν υπάρχουν αντιρρησει Ε, κυρία Κορνέλισεν. Η κυρία Κορνέλησεν θέλει το λόγο. Όχι, όχι. Άρα δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε με τη διευκρίνηση αυτή την ε, τροπολογία υπέρ, κατά. δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 5, άρχεται ψηφοφορία. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. 30 ε, με 27 η ε, τροπολογία η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίφθηκε τους, ε, αυτούς που δηλούσαν αποχή δεν τους λαμβάνουν υπόψη μας. Ε, το 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ, η ψηφοφορία, υπέρ 1, υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται και τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Chiusa la Κλείνει η ψηφοφορία. 49 υπέρ 7 κατά 3 αποχές άρα υπερψηφίζεται η εισήγηση με μεγάλη πλειοψηφία και τώρα έχουμε να ψηφίσουμε ε, το, την έκθεση σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα που προκύπτουν από την αστάθεια στόχος και ρόλος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η είναι ο κύριος Φιωρέλο Προβέ Λοιπόν, ε, τροπολογία 98. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, 100 με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές 101 ηλεκτρονικά ξεκινά λίγη 26 υπέρ, 30 κατά, 2 αποχές, άρα απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 107 ξεκινά λίγη εγκρίθηκε 31 υπέρ 26 κατά 108 υπέρ κατά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Λοιπόν, εντάξει. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 108. Αν αρχίσω εγώ να αμφιβάλλω... Λοιπόν, θα πρέπει να σεβαστείτε την ψήφο σας, οπότε 29 υπέρ 26 κατά άρα εγκρίθηκε συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στο 111 λοιπόν 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές, 115 ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινά. Ίσως έχετε κουραστεί να ε, ψηφίζετε και δεν σηκώνετε τα χέρια σας. 115 λοιπόν, λίγη ηλεκτρονική ψηφοφορία. 14 υπέρ, 41 κατά, απορρίπτεται. 117 υπέρ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 εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές 121 ε, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινάει Λίγοι 45 υπέρ 6 κατά βλέπετε δεν σηκώνετε καθόλου τα χέρια σας και 7 αποχές 130 υπέρ κατά αποχές μπράβο απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ όχι 136 Με συγχωρείτε, η 136 πρέπει να ψηφιστεί διότι δεν εγκρίθηκε η τροπολογία 130. Άρα 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερη συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 145 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία προφορική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία προφορική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 151 ξεκινάει. Λίγοι. Απερίφθη 51 κατά. Σας παρακαλώ τα χέρια σας είναι στις τσέπη σας. Η 152, ποιος είναι υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 153 υπέρ. Θέλετε την 152 να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ξεκινάει. Λίγοι. 32 κατά, 28 υπέρ, απορρίπτεται. Η 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 153 ξεκινάει η ψηφοφορία τώρα. Λίγη. 30 ε, κατά, ε, άρα απορρίπτεται υπέρ 28. 154 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα πάμε στην, ε, ε, στην 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 165 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε Θέλετε να ελέγξουμε την 166, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 166. Λίγη. 31 κατά, 29 υπέρ και απερίφθη. 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε τώρα συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 135, 35 ε, με συγχωρείτε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές για την 37 ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος λίγη εγκρίνεται 34 ψήφοι υπέρ 26 κατά 38 υπέρ κατά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 εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίφθη 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 49 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 50 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 52 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τώρα περνάμε στην 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθηκε. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 71 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 78 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές απερίπτεται. 87 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα Περνάμε στην τροπολογία 1 ή στα εκτιμώντας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά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 το 16 εφόσον εγκρίθηκε το 3 όχι άρα πάμε στο 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές άρα ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 18 τελειώνει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 18 εγκρίθηκε 25 κατά 36 υπέρ 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελευθεριών. Πρώτη τροπολογία, ε, λίμπε 1, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 2, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 3, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Λάμδα 4 ηλεκτρονικός έλεγχος της 3. Ξεκινάμε ηλεκτρονικό έλεγχο της ε, τροπολογίας 3 της Επιτροπής Ελευθεριών. Λίγη. «35 υπέρ, 24 κατά, εγκρίθηκε». Τώρα πάμε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 αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, τροπολογία 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Ε, ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία για το πρώτο μέρος της τροπολογίας 12. Λίγη. 29 υπέρ, 26 κατά, μία αποχή εγκρίθηκε. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, εντάξει δεν το θέλω Θέλετε να το ξαναδούμε. Ηλεκτρονική ως έλεγχος στις 15. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 15, λίγη, 28 κατά, 33 υπέρ, έχετε δίκιο, εγκρίθηκε. Δύο μέρη για την ε, τροπολογία 16. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 17 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γνωμοδότηση ΔΕΒΕ. Ε, πρώτη τροπολογία σε δύο τμήμα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο ε, μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία ελέγχου για την 3 υπέρ ε, ανοίγει λίγη 33 υπέρ 26 33 ε, ε, ε, κατά 26 υπέρ απερίφθη 4 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 8 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε να ελέγξουμε το δεύτερο μέρος ηλεκτρονικά ξεκινάμε Λίγοι. 36 υπέρ, 25 κατά, είχε σωστά εγκριθεί. Το 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ε, Καλυφτόμαστε από το άρθρο 50 και ξεχάσαμε την τροπολογία 28 όχι σε αυτό επί του 28 είναι η παρατήρηση. Πρέπει να ψηφίσουμε την 28, τροπολογία 28, την οποία ξεχάσαμε. Οπότε ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 28. Πηγαίνετε στη σελίδα 4 και θα δείτε ποια είναι η ένδειξη για την ψηφοφορία στην 28. Η Μπρίζα Τζικ που συνάδει με την συμβιβαστική 5 άρα ψηφίζουμε την 28 φαίνεται ασύμβατη αλλά είναι συμβατική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική, ε, τελικό ψήφισμα ε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινάμε λείπουν κάποιες ψήφοι, ορισμένα έχετε βάλει τις κάρτες χωρίς όμως να τα ακολουθήσετε και πρέπει με συγκίνηση να σας πω ότι ε, κέρδισε ο εισηγητής 53 υπέρ μία κατά και τρεις αποχές. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα την ε, τελευταία ε, ψηφοφορία που είναι η απαλλαγή του 2009 για το τρίτο τμήμα. Ε, η συγητής είναι η κυρία Ντεκάιζερ, τροπολογία υπαριθμών 1, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Οι δύο υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Οι τρία και αυτή απορρίφθηκε. Τέσσερα υπέρ, ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Η πέντε παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ε, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν η τελική ψηφοφορία. Έκλεισε. 53 υπέρ, ένα κατά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Ντεκάιζερ και ολοκληρώθηκε η, ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίε, η ώρα των ψηφοφοριών. Allora, invito, eh, il... Πρόεδρος, ε, καλό λοιπόν ε, τον ε, αντιπρόεδρο τον κύριο Πάσκο, τον κύριο Προβέρα, ένα από τους δύο να έρθουν εδώ να προεδρεύσουν γιατί προβλέπεται ότι θα παρουσιαστεί τώρα η δική μου εισήγηση. Eh, Ah, Colleagues, please, let's, let's move on and uh, start discussing uh, the annual report from the Council to the European Parliament. Λοιπόν, θα συζητήσουμε τώρα για την έκθεση του κυρίου Αλμπερτίνη. έκθεση του κυρίου Αλμπερτίνη. Και τώρα λοιπόν κύριε Αλμπερτίνη θα ήθελα παρακαλώ να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί θα ήθελα να αφήσω ε, τον απαραίτητο χρόνο στους συναδέλφους να σχολιάσουν ή να σχολιαστούν οι τροπολογίες τους. Αυτή λοιπόν η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας είναι η πρώτη που υποβάλλεται μετά τη σύσταση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ε, έχουμε 273 τροπολογίες, πολύ περισσότερες δηλαδή από εκείνες ε, που υποβάλλονται κατά κανόνα και αυτό λοιπόν υπογραμμίζει ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα ε, θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η νεοσυσταθήσα ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Βεβαίω ε, υπάρχει και μια σημαντική αναδιάρθρωση τη υπηρεσία αυτή. Σε αυτήν, εν πάση περιπτώσει, την έκθεση αναφέρεται για άλλη μια φορά ο καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, το οποίο μπορεί να είναι ένα όργανο ελέγχου και ε, καθορισμού κατεύθυνσης. Ε, οι τελευταίες εξελίξεις ε, κυρίως ε, στην Ανατολική Ευρώπη, στη Λευκορωσία, στη Μεσόγειο η ειδική αναφορά γίνεται για τις κρίσεις στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και στην Τινησία. Όλα αυτά καθιστούν απαραίτητο το κείμενο να προσαρμοστεί γιατί το κείμενο είχε συναχθεί πριν από κάποιες εβδομάδες. Πρέπει λοιπόν να λαμβάνει κανείς υπόψη του τις εξελίξεις και γι' αυτό ίσως είναι απαραίτητο να κατατεθούν και προφορικές τροπολογίες πριν λάβει χώρα η τελική ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ που θα λάβει χώρα στις 13 Απριλίου. Οι περισσότερες ε, τροπολογίες αφορούν την πολυμέρεια, τα Ηνωμένα Έθνη, τις διατλαντικές σχέσεις, το Κοσφοπέδιο, τη Ρωσία, την ε, Ανατολική Εταιρική Σχέση, την Αίγυπτο και την Τινησία. Εξάλλου, Υπάρχουν και κάποιες ε, άλλες συμβαστικές τροπολογίες που εξετάζονται για να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να περιοριστούν αυτές οι 273 ε, τροπολογίες προβλέπω να συζητήσω με τους ε, σκιώδης την εβδομάδα 28 έως 31 Μαρτίου. 25 είναι οι τροπολογίε υπό εξέταση και πρόκειται να καλύψουμε περίπου ε, τις ε, μισές από αυτές που έχουν κατατεθεί. Νομίζω λοιπόν ότι στις 12 Απριλίου πριν από την ψηφοφορία θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε στην Ολομέλεια τους τελικού συμβιβασμού. Υπάρχουν βέβαια κάποια επιχειρήματα, κάποια ποιες θέσεις ε, ε, για τις οποίες έχουν υποβληθεί περισσότερες τροπολίες και δεν θα τα μακρηγορήσω αλλά πρόκειται για τους γενικούς στόχους της πολιτικής ασφάλειας για την ε, συνεκτικότητα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης τη διαχείριση της κρίσης την πολιτική ενέργειας το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και κάποια άλλη ε, η σχέση με τον ΝΑΤΟ παρήματος χάρη δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σα αναφέρω όλους αυτούς τους τομείς γιατί μετά όταν θα συζητάμε τις συμβασίες τροπολογίε, έτσι και αλλιώ θα του δούμε αυτού του τομεί. Και υπάρχουν άλλε τροπολογίε για συγκεκριμένε γεωγραφικέ περιοχέ, τι οποίε και σα προανέφερα. Όπω ξέρετε, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται για τον Μάιο και στο σημείο αυτό ε, δεν έχω τίποτα άλλο να σα πω ε, και είμαι στη διάθεση των συναντέλφων ε, για να μα εξηγήσουν τι τροπολογίε του. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Σβόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο συνάλφος κύριος Αλμπερτίνη, ε, ο εισηγητής, μας επισήμανε τα βασικότερα θέματα και είπε βεβαίως ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι τελευταίες εξελίξεις. Κατ' ουσίαν πρόκειται για μια έκθεση που αφορά στο παρελθόν, την εξωτερική πολιτική του παρελθόντος. Νομίζω όμως ότι και κάποιες δικές μου αλλά και άλλες τροπολογίες καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο, στην έκθεση για το παρελθόν να συμπεριληφθούν και στρατηγικής φύσεως προτάσεις για το παρόν και για το μέλλον για αυτή τη χρονιά. Διότι de facto πλέον πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και στοιχεία τα οποία ε, δεν καλύπτονται από, την αρχική, από κάποια αρχική εισήγηση. Γι' αυτό λοιπόν τον πρόεδρο κύριο Αλμπερτίνη θα ήθελα να τον παρακαλέσω να συζητήσει με την ύπατη εκπρόσωπο μήπως ε, στο μέλλον μπορούμε εκθέσεις για το παρελθόν, σε εκθέσεις για το παρελθόν να περιλαμβάνεται και κάποιο κεφάλαιο για, την, για το τρέχον έτος ε, ίσως και για το μέλλον. Έτσι θα διευκολυνθεί κατά πολύ κατάσταση. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση και το επισήμανε αυτό ο κύριος Αλμπερτίνη αναφερόμεθα στο ρόλο της διπλωματικής υπηρεσίας και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης αξιολογούμε την υπηρεσία αυτή κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της. Δεν είναι εύκολο το καθήκον και θέλω να σας πω ότι με μεγάλη ανυπομονησία περιμένω ε, να δω πώς θα κρίνει την υπηρεσία αυτή ο κύριος Αλμπερτίνη, πώς θα κινηθεί μέσα σε αυτή την γάμα από θετικά μέχρι αρνητικά στοιχεία. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί αλλά και κάπω και διακριτικοί γιατί δεν έχει κανένα νόημα ε, στην Ολομέλεια σήμερα παραδείγματος χάρη στον κύριο Μπαρόζο να ασκούμε εντονότατη κριτική διότι ε, η κριτική αυτή ε, δεν ασκήθηκε μόνο από τους αντιπάλους αλλά και από άλλους. Η κυρία Άστρον βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά τα καθηκοντά της και πιστεύω όπως σας είπα μπορούμε σαφώς και να ασκήσουμε κάποια κριτική αλλά σε γενικές γραμμές η έκθεση αυτή θα πρέπει να στηρίξει το ρόλο της της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και όχι τόσο να επικρίνει γενικότερα το σύνολο της διπλωματικής υπηρεσίας. Αυτά που πρέπει να δούμε είναι και το πώς λειτουργήσαν οι διπλωματικές υπηρεσίες ε, τα τελευταία χρόνια, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι υπηρεσίες αυτές αντιμετώπισαν ε, πάρα πολλές δυσκολίες, ε, όχι ακριβώς αυτό το τεστ αντίστασης που ίσως πρέπει να γίνει στην Ιαπωνία αλλού, αλλά τεστ, στρες τεστ ήταν και αυτά. Μην ξεχνάτε τι έγινε στη Βόρεια Αφρική. Ε, είχαμε εκεί διπλωματικέ υπηρεσίε. Τι έγινε, βοήθησαν αυτέ. Απέκτησαν τι απαραίτητε πληροφορίε. Και έτσι φτάνω στο επόμενο σημείο. Εμεί δεν έχουμε μυστική υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καλό ίσω είναι αυτό, γιατί και να είχαμε τίποτα δεν θα έκαναν. Και αυτοί που είχαν, ε, τι κατάφεραν. Αλλά χρειαζόμαστε όμω ε, πληροφορία, υπηρεσία πληροφοριών που να συνεργάζεται με ΜΚΟ και με άλλου, κυρίω σε τέτοιου είδου καθεστώτα όπως αυτά που συναντάμε στη Βόρεια Αφρική, στον Κάφκαστο και στην Κεντρική Ασία. Πρέπει λοιπόν να αποκτάμε περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες από άλλους γιατί μπορούμε, με τον τρόπο θα μπορούμε να λειτουργήσουμε και καλύτερα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πώς μπορεί πράγματι να ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για καταστάσεις που διαδραματίζονται σε αυτές τις χώρες. Και φτάνω στο επόμενο θέμα, ε, στην ανατολική εταιρική σχέση. Εκεί λοιπόν έχουν κατατεθεί αρκετές τροπολογίες. Ήδη σήμερα είχαμε κάποιον, ε, κάποιες ψηφοφορίες, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι τελευταίες εξελίξεις. Και φτάνω στο τελευταίο σημείο της ε, παρέμβασής μου. Αναμφίβολα πρέπει να υπογραμμίσουμε, να στηρίξουμε περισσότερο τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά ας είμαστε ειλικρινεί όμως, οι επαναστάσεις στη Βόρεια Αφρική δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ξαφνική, τον ξαφνικό διακαή πόθο για τη δημοκρατία, αλλά και με την κοινωνική κατάσταση στην οποία έχουν περιπέσει πάρα πολλοί νέοι. Το γεγονός ότι δεν εκπληρώνονται πολλές από τις δικές τους προσδικίες και αυτό μέτρησε πάρα πολύ. Από τη μια οι άνθρωποι έχουν ε, καλή καλύτερη εκπαίδευση, όμως από την άλλη δεν έχουν θέση εργασία που ανταποκρίνεται στα προσόντα τους. Στο Ουσμπεκιστάν, παραδείγματο χάρη, επισκεφτήκαμε το Ουσμπεκιστάν και είδαμε εκεί πολλοί νέοι έχουν εκπαίδευση, αλλά δεν έχουν δουλειά. Ε, Ευτυχώ, ε, βέβαια, υπήρξαν ε, αυτέ οι αναταράξει και οι επαναστάσει, αλλά σα λέω, το θέμα δεν ήταν μόνο η δημοκρατία, ήταν και η κοινωνική δικαιοσύνη και βεβαίω και το περιβάλλον. Και αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν θέλω να αναφερθώ στην τραγική κατάσταση της Ιαπωνίας, αλλά ε, υπάρχουν και άλλα εξίσου δυσάρεστα. Κεντρική Ασία, Λιψιδρία, εχθές παραδείγματος χάρη. Ε, συζητήσαμε το θέμα της ανέγερσης ε, ενός μεγάλου υδατοφράχτη στο Τατζικιστάν που θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή. Αυτό λοιπόν ε, πρέπει να το λάβει υπόψη τη υπηρεσία εξωτερική δράση. και για αυτό το θέμα έχουν κατατεθεί πάρα πολλέ τροπολογίε. <clears throat> πρέπει να σα πω τελειώντας Κύριε Αλμπερτίνη, δεν σας ζηλεύω με όλο αυτόν τον αριθμό των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Εγώ εύχομαι, όπως σας είπα, να καταλήξουμε σε μια κοινώ αποδεκτή λύση, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε από τους άλλους ε, κοινή εξωτερική πολιτική και εμείς εδώ να είμαστε διχασμένοι. Εγώ προσωπικά έχω κάποιο πρόβλημα με την εβδομάδα 28 Μαρτίου, γιατί εμείς θα είμαστε στην Αθήνα με την πολιτική μου ομάδα. Ε, θα το δούμε, εντάξει, θα το δούμε σε διμερές επίπεδο. Πάντως, κατά τα άλλα, συμφωνώ να ψηφίσουμε στις 13 Απριλίου. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να επενθυμίσω στου συναδέλφου ότι στις 4.30 θα υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ε, τον Πρόεδρο. Δεν είμαι σίγουρος, λέει ο κύριος Πάσκο. Ο κύριος Νταφ. Α, οπότε θα πρέπει να είμαι ακόμη πιο σύντομος από ό,τι συνήθως. Είναι κάπως παράδοξο, κύριε Πρόεδρε, το ότι εξετάζουμε μια έκθεση που υποτίθεται ότι αφορά την εξωτερική πολιτική του 2009. Προμίας διετίας δηλαδή. Εγώ σχεδόν έχω ξεχάσει τι συνέβαινε στον κόσμο το 2009. Είχαμε εκλογέ, λέει ο κύριος Πάσκο. Ναι, αλλά Ίσως θα ήταν πιο λογικό να αναθεωρήσουμε τις διαδικασίες και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουμε τις αιτήσεις εκθέσεις. Να επιταχύνουμε κάπως το ρυθμό για να είναι πιο επίκαιρη η συζήτηση της αιτήσιας έκθεσης. Βέβαια, ήταν πραγματικά δύσκολη καιρή με την ίδρυση και θέση εφαρμογή της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και όπως είπε ο κύριος Φόποντα, καλό θα είναι να μην είμαστε υπερβολικά επικριτικοί με μια υπηρεσία που δεν έχει ακόμη πλήρως τεθεί σε εφαρμογή. Πάντως ο ρόλος της κάθε φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικός. Και μιλάω ως ένας από αυτούς που συνέβαλαν στην διατύπωση και προσδιορισμό των εξουσιών του είπατε εκπροσώπου κατά την σύνταξη της συνθήκης. Και είναι πραγματικά περίπλοκο το πλέγμα ευθυνών και αρμοδιοτήτων της είπα της εκπροσώπου. Εγώ γενικώ ε, την υποστηρίζω, αλλά νομίζω ότι πολύ συχνά θεωρεί τον εαυτό της ως το μεσάζοντα μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής και δεν ε, συμπεριφέρεται ως ε, συνήγορος υπέρμαχος ε, της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας γιατί με βάση την ε, συνθήκη έχει την ε, αρμοδιότητα και την εξουσία να προτείνει κοινή πολιτική. Πολύ συχνά όμως δεν καταφέρνει να επιτελέσει αυτό το σκόπο. Και σε ό,τι αφορά την τροπολογία στην παράγραφο 4, προσπάθησα εκεί να παρουσιάσω όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της που ξεκινάει από την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ε, εξωτερική πολιτική και την εφαρμογή περνώντας από την εφαρμογή και καταλήγοντας στην ε, συμμόρφωση των κρατών μελών στο Συμβούλιο υπάρχει διαφωνία μεταξύ των κρατών μελών για θεμελιώδη ζητήματα. Γνωρίζουμε ποια είναι τα προφανή. Το Κωσυφοπαίδιο, η Μακεδονία, η Τουρκία. Υπάρχουν όμως και καμουφλαρισμένες διαφωνίες ή συγκεκαλυμμένες διαστάσεις απόψεων ή αντίθετες απόψεις μεταξύ κρατών μελών που έχουν και ιστορικές διαστάσεις. Και αυτό είναι μερικές φορές δύσκολο να γίνει λεπτό. Πάντως, εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε μια διαφωνία και να τις φέρουμε στο φως προσπαθώντας να διαλευκάνουμε το σκο... τις αιτίε αυτών των διαφωνιών. Αν δεν γίνει μια τέτοια διεξοδική ανάλυση δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση. Και νομίζω ότι του χρόνου ένα θεμελιώδες ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η Τουρκία. Γιατί νομίζω ότι έχει καταρρεύσει η στρατηγική μας για την Τουρκία. Ακόμη και η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας έχει αποτελματωθεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να, δεχόμαστε διαμαρτύρητα την απώλεια της Τουρκίας από την ευρωπαϊκή σφαίρα επιρροής. Και η Τουρκία είναι πολύ θορυβημένη με την όλο και μεγαλύτερη απόκλησή της πια από την ενταξιακή προοπτική. Κάτι άλλο που θα πρέπει να προωθήσουμε είναι διακοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων στα θέματα ΚΕΠΑ και κοινή πολιτικής άμυνας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολες. και υπάρχουν ακόμη πολλές παρεξηγήσεις και παρανοήσεις στα εθνικά κοινοβούλια σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα ε, και τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το πλήρες φάσμα της διεθνούς πολιτικής. Και ελπίζω ότι η Επιτροπή μας θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα αυτό. Φαντάζομαι θέλετε να σταματήσω εδώ και αυτό θα κάνω. Πω, διαβάσε το μυαλό μου. Μπράβο. Ο κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ. Όπως ξέρει ο κύριος Αλμπερτίνη, γιατί κατά την αρχή της συζήτησης είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, ε, η ομάδα μου δεν θα καταψηφίσει την έκθεση, αλλά θα υποβάλει μια έκθεση μειοψηφία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ε, συμφωνούμε με την κρατούσα άποψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για θέματα ασφάλεια, ούτε για θέματα εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρω ε, οι μεγαλύτερε ομάδε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι καλό θα ήταν να κάνω μια αναθεώρηση και ίσως τα θέματα ασφάλειας να τα στηρίξουμε σε μια αποτροπή με βάση το διατλαντικό μας ε, σύνδεσμο και το ΝΑΤΟ που είναι ένα πείθμενο πηγάδι με πολιτικές βιομηχανικές διαστάσεις και μάλιστα έχουμε τεράστιες δαπάνες και το ενώ το πηγάδι του ΝΑΤΟ γίνεται απίθμενο, το πηγάδι των, ε, των στόχων της χιλιετίας ε, έχει στερέψει. Έχουμε πολύ πιο αξι... αξιόλογους στόχους την εκρίζωση της φτώχειας, την περιθωριοποίηση, γιατί με την ανισότητα τη λιμοκτονία, την ε, εξαθλίωση. Αυτά είναι που... Αυτοί οι λόγοι είναι που δημιουργούν τεράστια όπλα και δημιουργούν τεράστια ανασφάλεια. Ούτε πιστεύω ότι θα ήταν καλό αυτή τη στιγμή τον 21ο αιώνα να προσκαλέσουμε τα κράτη-μέλη να αναπτύσσουν ε, τις στρατιωτικές τους δυνάμεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου ξεπερνώντας τα εθνικά του σύνορα. Αυτό κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε βέβαια και τηρούν αυτή την πολιτική αποτροπή του ΝΑΤΟ. Αλλά δεν συμφωνώ με κάτι τέτοιο, γιατί και εκείνα θα είχε το δικαίωμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν αυτός ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ανασφάλεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Η πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει απογυμνωθεί στα πλαίσια της εξωτερικής μας πολιτικής. Δεν είναι ότι οι μυστικές υπηρεσίες δεν ήξεραν τι συνέβαινε στην Τινησία, στην Αίγυπτο ή στη Λιβύη. Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες στις κεντρικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το θέμα είναι ότι ο προσανατολισμός της ε, ε πολιτικής γειτονίας συνεργάστηκαν με τον Μπεναλή, τον Μουμπάρα και τον Καντάφη. Ήμασταν συνεργάτες, συνένοχοι. Συνεργαστήκαμε και παρά τις συμφωνίες σύνδεσης που είχαμε, όχι με τη Λιβύη βέβαια, παρόλο που είχαμε διαπραγματεύσεις. Είχαμε όμως συμφωνίες σύνδεση με την Αίγυπτο και την Ισία. Και αυτές οι συμφωνίες σύνδεσης είχαν το άρθρο 2 για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Και όμως δεν τηρήθηκε ποτέ, δεν εφαρμόστηκε ποτέ αυτό το άρθρο. Το ίδιο γίνεται και με τον Νατανιάχου. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το Ισραήλ. Οπότε καλό θα ήταν κυρίες και κύριοι να έρθει μια στιγμή που θα να σκεφτούμε σοβαρά μήπως χρειάζεται να επαναπροσανατολίσουμε την εξωτερική μας πολιτική και την πολιτική μας ασφάλειας και άμυνας. Γιατί η κατάσταση που βιώνουμε τώρα στη Βόρεια Αφρική μας ε, δείχνει ότι μάλλον κάπου κάναμε λάθος και ίσως θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε και το θέμα του επαναπροσανατολισμού της εξωτερικής μας πολιτικής. Κύριε Αλμπερτίνη, μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια αναθεώρηση για να φτάσουμε σε ένα σύστημα ασφάλειας που θα επιδιώκει στόχους όπως ο αφοπλισμός και να βάλουμε την πολιτική πάνω από οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Τα Ηνωμένα Έθνη και αναθεωρημένα Ηνωμένα Έθνη είναι κάτι που απαιτεί ο 21 ο αιώνα, ώστε πραγματικά να γίνουν τα Ηνωμένα Έθνη η κυβέρνηση του κόσμου και κανείς δεν μπορεί να παραγωνίζει τα Ηνωμένα Έθνη και να ε, δρά μέρο. Μου δείχνετε το ρολόι κύριε Πρόεδρε. Πάντω πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα πολύ άμεσο πρόβλημα που είναι η στρατιωτική κατοχή τη Τουρκία με 40.000 ε, στρατιώτε ε, στο βόρειο τμήμα τη ε, δημοκρατία τη Κύπρου που είναι μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι αυτό χρήζει πολιτική, διπλωματική δράση και ε, στεναρής ενέργειας και εγχειρήματο και να πούμε στην Τουρκία ότι είναι απαράδεκτη αυτή η πολιτική κατοχή που ασκεί στην Κύπρο γιατί έτσι... Ε, δίνει, προωθεί την απεικιοκρατοποίηση εκ μέρου των τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει ε, η Τουρκία επιτρέποντας αυτή την απεικιοκρατία και θα πρέπει να πούμε στην Τουρκία ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή την πολιτική γιατί έτσι αμφισβητεί την ε, ίδια την ταυτότητα του λαού των τουρκοκυπρίων. Η κυρία Λούνατσεκ και προσοχή στο ρολόι. θα ήθελα να επικεντρωθώ σε διάφορα θέματα τα οποία έχουμε, ε, στα οποία έχουμε προτείνει τροπολογίες για να συμπεριληφθούν στο ψήφισμα. Το ένα είναι αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο κύριος Νταφ, δηλαδή ε, το τι θέλουμε από την κυρία Άστον που λειτουργεί σαν υπουργό Εξωτερικών μας και συμφωνώ με τον κύριο Νταφ ότι περιμέναμε από αυτήν να είναι περισσότερο κινητή κινητήρια δύναμη στις εξωτερικές υποθέσεις και αυτό είναι στην εντολή που έχει λάβει. Μπορεί να το πράξει. Άρα πρέπει να τις διευκρινίσουμε ότι τη στηρίζουμε. Πρέπει να προχωρήσει έτσι ακόμη και αν όλα τα κράτη-μέλη δεν τις δίδουν αυτή τη στήριξη θα έπρεπε να θεωρήσει ότι η δικιά μας στήριξη είναι σημαντική εις τη λειτουργία των αρμοδιοτήτων της και είναι είναι ένα ουσιαστικό μέρος από αυτά τα οποία περιμένουμε να κάνει. Ένα άλλο που πρέπει να ενισχύσουμε είναι ε, η ε, μεσολάβηση για τις ε, διαφορές για την ESP, για CSDP και εκεί έχουμε μια τροπολογία μαζί με άλλες ομάδες οι οποίες ζητούν από την κυρία Άστον να βασιστεί στην δήλωση που είχε κάνει πέρυσι τον Ιούλιο ότι θα συμβάλλει στην εγκαθίδρυση Ειρήνη. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ένα Συμβούλιο εκπαιρεώσεως Κρίσεων με ε, αυτή την εντολή να προλαβαίνει τις ε, διαφορές και να επιλύει τις ε, διενέξεις. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα θέλαμε να ζητήσουμε είναι να αντιπαρέλθουμε τη την, ε, ε, ε, την, τις δυνατότητες διότι υπάρχουν πολλοί που εμπλέκονται και οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί και θα πρέπει να στηρίξουμε τους πολιτικούς και τους πολίτες ελάχιστη είναι η κοινή μικτή οργανισμοί που είναι και και στρατιωτικοί και εκπρόσωποι των πολιτών. Οπότε, ε, πρωτού φτάσω στο τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι κάναμε μια συζήτηση για το ΝΑΤΟ, ότι ε, ε, θεωρήσαμε ότι καλό θα ήταν να πούμε στην έκθεσή μας ότι λυπούμεθα που δεν προχωρήσαμε στον πυρηνικό αφοπλισμό και ε, να υπάρχει επίσης ε, ε, μια δυνατότητα επιλύσεως κρίσεων που θα έπρεπε να έχει γίνει και με, σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Στη Συμφωνία της Θεσσαλονίκης το 2003 είχαμε συμφωνήσει ότι στόχος μας είναι όλες οι χώρες των Βαλκανίων να περιληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να ξεκινάμε, ξεκινήσουμε αμέσως στον διάλογο των θεωρήσεων με το κοσυφοπαίδιο. Ευχαριστώ. Όσοι μίλησαν και παρενέβησαν μέχρι στιγμής ήταν σκιώδεις εισηγητές, γι' αυτό τους δώσαμε περισσότερο χρόνο. Έχουμε άλλους δύο μιλητές τώρα και θα παρακαλούσα να περιοριστούν σε δύο λεπτά ο καθένας. Η κυρία Μουνής καταρχήν και ο κύριος Μιλανμόν μετά. Ευχαριστώ. Η ετήσια έκθεση είναι πολύ σημαντική γιατί διαμορφώνει ένα δόγμα της Επιτροπής Εξωτερικών και περιλαμβάνει αυτά που έχουμε εγκρίνει και σε προηγούμενες εκθέσεις, όχι μόνο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που είναι το έτος αναφοράς της ετήσιας έκθεσης, γιατί θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το χρονικό ορίζοντα για να μην είμαστε πια παροχημένοι, αλλά ακριβώς επειδή προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα δόγμα και μια στάση συνεπή, έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά το κοσυφοπαίδιο, ειδικά σε αυτή την έκθεση, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση σε ό,τι αφορά την επίσημη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά που λέμε για το κοσυφοπαίδιο θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την επίσημη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κοσυφοπαίδιο. Επίσης, ό,τι αφορά τους μηχανισμούς της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, του, τους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς και τα μέσα, αυτά θα πρέπει να αναφέρονται και στις φιλοδοξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχει στην, στον έλεγχο της εφαρμογής των διαφόρων μέσων. Για παράδειγμα, έχουμε το μέσο σταθερότητας που βρίσκεται σε ένα νομικό λίμπο αυτή τη στιγμή, σε μια σε ένα νομικό κενό και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει τις αρμοδιότητες που κατοχυρώνονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχω μια τροπολογία για την Αίγυπτο επίσης, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο εισηγητής θα πρέπει να καταθέσει προφορικές τροπολογίες για τις υπόλοιπες χώρες στις οποίες είχαμε τέτοια περιστατικά και διαμαρτυρίες ή διεκδικήσεις αλλαγής. Νομίζω ότι υπάρχει πια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά αυτές τις μεταβατικές ε, αρχές. Για το Ιράν θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη διατύπωση και να ευθυγραμμιστούμε με αυτά που ψηφίσαμε στην έκθεση Μπέλντερ. Το ίδιο και για τη Μέση Ανατολή. Και προκειμένου να επικαιροποιήσουμε την έκθεση, καλό θα ήταν να αναφερθούμε και στο θέμα του Σουδάν και στην έκβαση του δημοψηφίσματος στο Σουδάν. Αυτά δεν θα μακρηγορήσω. Αυτά είχα να πω για τις τροπολογίες μου. Σας ευχαριστώ κύριε Σμιγιαρμόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα με δυο λόγια να συγχαρώ τον κύριο Αλμπερτίνη για την έκθεσή του, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ πλήρης, οριζόντια, ισορροπημένη και μεστή έκθεση και ίσως το μόνο της ελάττωμα, αν είναι να βρούμε κάποιο, είναι η ημερομηνία της, γιατί δεν έλαβε υπόψη τη, τα, συμβάντα στην Αίγυπτο και στις υπόλοιπες χώρες του Μαγκρέπ. Γι' αυτό και κατέθεσα κάποιες τροπολογίες ίσονο σημασία, προκειμένου να επικαιροποιήσουμε αυτό το τμήμα της ε, έκθεσης ε, για τα περιστατικά στην νότια όχθη της Μεσογείου. Και όπως είπε και η κυρία Μουνής, και εγώ θα ήθελα να αναφερθούμε αφέστερα προς το κοσυφοπέδιο, ώστε να είναι αντιπροσωπευτική έκθεση και να μην λαμβάνει υπόψη μόνο τη θέση 5 από τις 27 χώρες ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αναγνώρισαν ε, την ανεξαρτησία του κοσυφοπεδίου. Αυτά επαναλαμβάνοντας τις ευχαριστήσεις και τα συγχαρητήριά μου προς τον κύριο Αλμπερτίνη. Ελπίζω να συνεχίσει με το διαλλακτικό, γενναιόδωρο και ανοιχτό του πνεύμα και να συμπεριλάβει και αυτές τις τροπολογίες στην έκθεσή του. Σας ευχαριστώ. Έχει καταφτάσει όπως και κλειμένος μας και ξέρετε ότι θα πρέπει να ακούσουμε και τις απαντήσεις του κύριου Αλμπερτίνη στα σχόλιά σας. Γι' αυτό είμαι από τον κύριο Παπόφσκι που δεν θα του δώσω το λόγο, αλλά προτιμώ να δώσω το λόγο στον κύριο Αλμπερτίνη για να σχολιάσει αυτά που ακούσαμε από τους συναδέλφους. Όπως ε, σας είπα ήδη, οι παρατηρήσεις που ακούστηκαν εδώ και που τις άκουσα και εγώ, όλες αυτές οι παρατηρήσεις είναι ιδιαίτερα εύστοχες, κυρίως αυτές που αναφέρονται στην, στις ταχύες, ταχύτατες εξελίξεις, κάποιες, ε, κάποιους αστάθμιτους παράγοντες στη διεθνή σκακέρα, τόσο στην ε, Μεσόγειο όσο και στην στις ανατολικές ε, περιοχές Ευρώπης. Μιλάμε για καταστάσεις που εξελίχθηκαν ανώμαλα και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να υπάρξει διόρθωση της έκθεσης, κάτι το οποίο θα το λάβω υπόψη μου. Όσα λοιπόν ελέγχθησαν σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου, αλλά και με την ε, πραγματοποίηση, την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής, όλα αυτά θα τα αξιολογήσω ιδιαίτερα και θα δείτε ότι αυτά θα τα παρουσιάσω και στις συμβαστικές προτάσεις που θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, ε, ε, δεν θα μακρηγορήσω, θα μιλήσω μόνο για ένα ακόμα λεπτό για να είμαστε πραγματικά ακριβείς στο χρόνο που θα υποδεχθούμε τον προσκεκλημένο μας υπάρχουν οι προφορικές τροπολογίες για να είναι πιο, επίκαιρες, ε, η, πιο επίκαιρη έκθεση αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ στην έκθεση αυτή γίνεται λόγος ε, για τον προηγούμενο χρόνο και ας μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκαν πάρα πολλές αναταράξεις ε, και πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα ε, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη μας επιχειρήματα ε, τα οποία ε, είναι ακόμα και πιο παλιά. Αυτό βέβαια δεν μας αφαιρεί τη δυνατότητα να εξετάσουμε το τι ακριβώς συνέβη και να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Θέλω να σας πω ότι εγώ βεβαίως και είμαι στη διάθεσή σας για να λάβω υπόψη μου τις συμβαστικές τροπολογίες και θα θελήσω να ε, ακούσω και τα σχόλιά σας όλα εκείνα τα οποία είχατε ήδη την ευκαιρία να το κάνετε. Όσα είπατε θα δείτε ότι θα αντικατοπτρίζονται στις συμβαστικές τροπολογίες. Ε, σας ευχαριστώ και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ας ε, προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Ας συνεχιστεί η σημερινή συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον ε, προσκεκλημένο μας να έρθει εδώ μπροστά στο Προεδρείο για να ε, ξεκινήσουν οι εργασίες. Πολύ ωραία λοιπόν. Ας ε, καλωσορίσουμε τον ε, Πρωθυπουργό της Αρμενίας, ε, τον κύριο Τιγκράν Σαργζιάν. Ελπίζω να μην κατακρεούργησα το όνομά σας. Ο Πρωθυπουργό της Αρμενίας μας κάνει την τιμή να μας, επισκεφθεί. Θα ήθελα λοιπόν να τον καλωσορίσω και θα ήθελα να καλωσορίσω, ε, θα ήθελα να είχα μπορέσει να καλωσορίσω τον πρώτο αντιπροσωπή στην Αρμενία, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν είναι παρόν και γι' αυτό δεν μπορώ. Ε, για μας η δική σας επίσκεψη κύριε ε, Πρωθυπουργέ είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις με την Αρμενία. Οι σχέσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο φάσμα σχέσεων μέσα ε, στο πλαίσιο της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ε, γειτονίας, η οποία είναι μια πολιτική που βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης. Στις 20 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της πολιτικής και η δική μας Επιτροπή σήμερα το πρωί ψήφισε σε ένα κείμενο που αφορά ακριβώς αυτή την πολιτική γειτονίας και επαναλαμβάνω ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί άπτεται των ε, παγκόσμιων και διεθνών σχέσεων. Εμείς ε, λοιπόν ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την ε, ανατολική εταιρική σχέση. Αυτήν την πολιτική την θεωρούμε ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για, την, για τον εξυγχρονισμό των χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την διαδικασία εκδημοκρατισμού στη Μεσόγειο και με τον ίδιο τρόπο θεωρούμε ότι η πολιτική γειτονία και αυτή έχει ως στόχο να προάγει τις δημοκρατικές αρχές στις γειτονικέ μας χώρες. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, και στη δική σας τη χώρα πρόσφατα έλαβαν χώρα διαδηλώσεις που οργανώθηκαν από την αντιπολίτευση. Ε, ίσως ε, μου επιτρέπετε να προτάξω ε, ή να προτρέχω με κάποιες ερωτήσεις που θα υποβάλουν οι συνάλφοι. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε για την φύση αυτών των διαδηλώσεων. Πώς σκέπτεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτές τις διαδηλώσεις. Εμείς θέλουμε να υπάρχει θετικός διάλογος, να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των αντιφρονούντων, να γίνονται σεβαστοί οι δημοκρατικοί κανόνες. Τέλος, ένα επιχείρημα τελευταίο, εξίσου σημαντικό αφορά στην ε, διένεξη στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Το Κοινοβούλιο ανέκαθεν προσπαθούσε να, να εφαρμόσει ε, μία ε, πολιτική διαμεσολάβησης Δηλαδή επιβεβαιώνουμε ε, τις αρχές του Μίνσκ, την δήλωση της Μόσχας, ε, της Μαδρίτης, όλα δηλαδή ε, αυτά τα θέματα και πολιτικές που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο, ένα έγγραφο το οποίο εμείς στηρίζουμε και θεωρούμε ότι οι κυβερνήσει τη Αρμενία και του Αζερβαϊτζάν θα πρέπει να καταλήξουν σε μια ειρηνική διευθέτηση του προβλήματο. Ε, νομίζω ότι σα αφαίρεσα κάποιο χρόνο. Ε, είπα ήδη πολλά. Δεν θα σα αφαιρέσω περαιτέρω το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σα. Περιμένουμε να ακούσουμε τι απόψει σα ε, και θα διεξεχθεί συζήτηση περίπου μέχρι τι 5.30 το απόγευμα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, βέβαια μπορείτε να αρχίσετε το χρόνο σας ε, όπως θέλετε, αλλά θα έλεγα καλύτερα θα ήταν να μην ξεπεράσετε τα 10 με 15 λεπτά. Το λόγο έχετε εσείς κύριε Πρωθυπουργέ. Dear Mr. Albertini. Αγαπητέ κύριε Αλβερτίνη, ε, πρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Έχω, νιώθω μεγάλη τιμή σήμερα που απευθύνομαι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας ευχαριστώ που διοργανώσετε αυτή τη συνάντηση. Ό,τι θέματα είναι σήμερα στην ημερήσια διάταξη πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια των προσφάτων εξελίξεων ε, παγκοσμίω. Τι υποκινεί την ε, τρέχουσα, τις τρέχουσες ταραχές ε, κρίσης και διενέξεις στη Μέσο Ανατολή και Βόρειο Αφρική. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο κόσμος θέλει αλλαγή. Ξέρουμε όμως από την ιστορία ότι όλες οι ιστορίες δεν καταλήγουν στον επιζητούμενο στόχο και γι' αυτό πιστεύω ότι η επιτυχία των ουσιαστικών αλλαγών εξαρτάται από τη δυνατότητα να διατυπώσουν συλλογικά στόχους και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του λαού στη διαδικασία επιτυχίας τους η πείρα των ευρωπαϊκών κρατών αποδεικνύει σαφώς την αποτελεσματικότητα των δημοκρατικών ε, θεσμών στην επίτευξή τους και συγχρόνως σέβεται το βασικό δικαίωμα ελευθερίας εκφράσεως και τη σημασία του πλουραλισμού και δημοσίας συζητήσεως. Η Αρμενία πάντοτε έχει ε, συνειδητά επιλέξει την ευρωπαϊκή οδό ανάπτυξης. Ο στόχος μας και η επιλογή μας προέρχεται από τις κοινέ χριστιανικές ρίζες της κληρονομιάς μας και την απόφαση να απομακρυνθούμε από το παρελθόν των αυτοκρατικών καθεστώτων. Η κληρονομιά της ε, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Σοβιετικής Ενώσεως έχουν επηρεάσει την κοινωνική μας συμπεριφορά αλλά οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις αρχίζουν να ε, παρουσιάζουν αποτελέσματα και να βελτιώνουν την ε, εκλογική διαδικασία, να ενισχύουν την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, να εξασφαλίζουν την ε, ανεξαρτησία ε, της δικαιοσύνης και να προωθούν την παρουσία μίας μέσης τάξης η οποία να είναι οικονομικά και κοινωνικά υπεύθυνη ψηφοφόροι και πολίτες αλλά σήμερα οι αλλαγές είναι πάρα πολύ ραγδαίες. Γι' αυτό και η Αρμενία πρέπει να επιταχύνει την εφαρμογή των αλλαγών και των θεσμικών μετατροπών διότι ε, είναι σαφές ότι τεχνική βοήθεια και η οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι σημαντικότατη για να έχουμε γρήγορη και ουσιαστική πρόοδο. Στα πλαίσια αυτά η ανατολική εταιρική σχέση που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα βασικό μέσων για να προωθηθεί η διαδικασία αλλαγής και επαναλαμβάνουμε την ευγνωμοσύνη μας για την προσφορά και την ε, πρόθεσή μας να αναπτύξουμε σύντομα την οικονομική και πολιτική μας ένταξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, διαπραγματευόμαστε μία συμφωνία συνδέσεως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούμε να ξεκινήσουμε συζητήσεις για μία ουσιαστική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Ένωση. Χάρη στη βοήθειά σας έχουμε μπορέσει ήδη να εφαρμόσουμε ένα ισχυρό γραφείο συνηγόρου του του πολίτη στην Αρμενία και μια διπλωματική σχολή. Ε, υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις δομές της αρμενικής κυβερνήσεως και ένα ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Δύο άλλα βασικά θέματα είναι η στήριξη των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη και η στήριξη της πρόσβασης στη δικαιοσύνη στην Αρμενία που είναι εν εξελίξει αυτή την εποχή και κατά αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ε, οικονομική και ε, δικαστική αναμόρφωση στην ε, Αρμενία. Το ε, αρνητικό είναι ότι υπάρχουν ε, διάφοροι κίνδυνοι γεωπολιτικοί στην περιοχή του Νοτιού Καυκάσου και καταρχάς η ε, εχθρική ρητορική του Αζερμπανιτζάν και ιδιαίτερος η επιθυμία να λύσει το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ πολεμικών μέσων εντείνοντας τις πολιτικές εντάσεις της περιοχής και δεύτερον, ο συνεχής αποκλεισμός της Αρμενίας από την Τουρκία μειώνει τις δυνατότητές μας να διαφοροποιήσουμε την οικονομία μας και οι φιλοδοξίες της Τουρκίας επηρεάζουν αρνητικά στην περιοχή μας τις ειρηνευτικές συζητήσεις για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Τέλος, χωρίς πρόθεση να ε, ε, να αμφισβητήσουμε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ενώσεως να διατηρήσει την ειρήνη θέλω να τονίσω ότι το γεγονός ότι υπάρχουν διεθνείς κυρώσεις εναντίον του Ιράν θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας οικονομικής αναπτύξεως διότι η μόνη διέλευσή μας είναι μέσω της γεωργίας και τα τραγικά γεγονότα της περιοχής τον Αύγουστο του 2008 απέδειξαν <clears throat> τον ευάλωτο χαρακτήρα της αρμενικανικής οικονομίας που οφείλεται στην υπερβολική εξάρτηση από ένα μοναδικό διάδρομο μεταφορών. Τότε μπορούσαμε να οργανώσουμε τις μεταφορές των βασικών πρώτων υλών μέσω του Ιράν. Αλλά η ε, επιδίνωση των κυρώσεων μείωσε αυτή τη δυνατότητα ε, και γι' αυτό έχουν, ε, και μεταξύ έχουν αποτύχει και οι συζητήσεις ε, και κοινές προσπάθειες με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξουμε ε, τα σύνορα της Τουρκίας. Γι' αυτό και οι λανθάνουσες διαφορές που υπάρχουν στον Νότιο Κάφκασο μπορούν να μειωθούν μόνο με μία κοινή πλατφόρμα αξιών και ευρωπαϊκή οδό προς την πρόοδο. Αναγνωρίζουμε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα συμβάλλουν στην ασφάλεια και συνεργασία της περιοχής και η μόνη βιώσιμη εναλλακτική λύση για τις χώρες της περιοχής μας πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στην ανοχή και στην αλληλεγγύη οι οποίες είναι οι ακρογωνιές λύθη της, σύντομη, της σύγχρονης Ευρώπης. Η κρίση απέδειξε τα ουσιαστικά προβλήματα της χώρας μας, ανεπαρκής διαφοροποίηση της οικονομίας, ανεπαρκές σύστημα δημοσίας διοικήσεως και, μία, και συνθήκες ανταγωνισμού. Επιπλέον η οικονομική κρίση οδήγησε σε μια μεγαλύτερη φτώχεια και μια αύξηση του εξωτερικού δημοσίου χρέους και υψηλό πληθωρισμό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν μειώσει τη δυνατότητά μας να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να επιλύσουμε τα προβλήματα που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Συνάδελφοι, τώρα θέλω να παρουσιάσω το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα σε θεσμικά θέματα με, λίγα λόγια. Η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η ύπαρξη ε, ισχυρών δημοκρατικών θεσμών, μιας ε, δραστήριας κοινωνίας των πολιτών, ελεύθερια εκφράσεως και ε, δίκαια εκπροσώπηση είναι βασικά για να να υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Επίσης μη ε, ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα εξασφαλίσει τα δημοκρατικά δικαιώματα. Η παιδεία μπορεί επίσης να αυξήσει τις δυνατότητές μας και μία σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς σύγχρονα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ισότητα για την οικονομία αγοράς που θα λειτουργεί σωστά και δεν είναι δυνατό να υπάρξει ανταγωνισμός χωρίς μεταρρυθμίσεις στη φορολογία και στους δασμούς. Η διαφθορά και η ανεπαρκής δημόσια διοίκηση είναι σοβαρά προβλήματα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων γι' αυτό και έχουμε υιοθετήσει ένα πρόγραμμα ενάντια στη διαφθορά και αυτή τη στιγμή δημιουργούμε τη σχετική νομοθεσία πέραν αυτού θέλουμε να έχουμε καλό σύστημα υγιεινής, να μειώσουμε την φτώχεια και να βελτιώσουμε το σύστημα συντάξεων. Θέλουμε να ενισχύσουμε και την εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή μας, το οποίο θα επιτύχουμε μόνο αν τα μέτρα που παίρνουμε είναι αποτελεσματικά. Είμαι βέβαιος ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι ουσιαστική για την Αρμενία για να επιτύχει προς αυτή την κατεύθυνση και θα μας δώσει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τους κινδύνους και να εξασφαλίσουμε μακροοικονομική σταθερότητα. Συνοψίζοντας η τωρινή μας κατάσταση χρειάζεται ριζικές αλλαγές και ε, τολμηρές πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα βασικό ρόλο για να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Νότιο Κάφκασο μέσω πιο δραστήριας εμπλοκής στην περιοχή και μεταρρυθμίσεων. Η Αρμενία χρειάζεται τη στήριξη των δωρητών για να καλύψει τα κενά μεταξύ των ε, δυνατοτήτων μας μεταρρύθμισης και των δεδηλωμένων αξιών μας και με την ηγεσία του Προέδρου η Αρμενία μπορεί να ε, επιταχύνει τις, ε, τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και είμαστε δεσμευμένοι για μια αποδοτική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις θέλετε να μου απευθύνετε. Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ. Ο πρώτος ε, που θα λάβει το λόγο είναι ο κύριος Βίγνη που είναι ο ε, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ε, Euronest. Είναι ο κύριος Βιγγένιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων κύριε Πρωθυπουργέ. Οι πληροφορίες που μας δώσατε είναι πολύ σημαντικές και αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι η δύσκολη κατάσταση φυσικά που αντιμετωπίζει η Αρμενία. Αυτό μας συγκλονίζει γιατί έχει τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στη χώρα. Για μερικά από τα προβλήματά σας ε, επαφίεστε στη διεθνή βοήθεια. Ούτε η χώρα σας ούτε εσείς προσωπικά δεν μπορείτε να βελτιώσετε για παράδειγμα τη σχέση σας με το Ιράν γιατί δεν έχετε κανέναν έλεγχο Ε, στα θέματα της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στη χώρα αυτή, αλλά θα μπορούσατε να έχετε κάποιο αντίκτυπο σε ένα άλλο φλέγο θέμα, ίσως το πλέον φλέγο θέμα για σας, που είναι η, η σύγκρουση στον Αγκόνο Καραμπάχ. Και από την άποψη αυτή θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας πώς εξηγείτε την έλλειψη πρόοδου στις διαπραγματεύσεις για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και υπάρχουν όλο και περισσότερες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Και αυτό ισχύει για κάθε σύγκρουση. Όταν δεν υπάρχει πρόοδος, δεν φταίει ποτέ μόνο η μία πλευρά. Πιστεύετε ότι η χώρα σας, η Αρμενία, μπορεί να προσφέρει κάτι ακόμη ή μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποια από τα λάθη που διαπράξατε μέχρι στιγμής. Και παρά τη δυσχερή κατάσταση, προοπτικές σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας είναι πολύ καλές, πολύ θετικές και ευνοϊκές. Η Συμφωνία Σύνδεσης θα βοηθήσει την Αρμενία να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν ή ε, διαπραγματεύσει για μια βαθιά εμπορική σχέση ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα σας ευνοήσει. Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες αυτές, ποιες είναι οι σχέσεις σας με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά την Τελωνιακή Ένωση. Σας έχει κάνει μια προσφορά η Ρωσία για πιθανή συμπερίληψη της Αρμενίας στην Τελωνιακή Ένωση μεταξύ Ρωσίας, Καζακστάν, Λευκορωσίας και από ό,τι ξέρω έγινε προσφορά για ένταξη στην Τελωνιακή Ένωση και σε άλλες χώρες. Ή μήπως πιστεύετε ότι αυτή η δυνατότητα αντιβαίνει στην ε, Συμφωνία ε, Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τις διευκολύνσεις για τις θεωρήσεις, άκουσα ότι ο κ. Μπαρόζος σας έδωσε κάποια θαρρυντικά μηνύματα για το θέμα των θεωρήσεων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της ε, άμεσης έναρξης των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό, ώστε να μπορέσουν οι Αρμένοι να επισκέπτονται ελεύθερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ως επικεφαλής της αντιπροσωπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωνές θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοδομητική θέση που είχε μέχρι στιγμής η Αρμενία για το θέμα αυτό και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα και μέσα σε ένα μήνα θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε την Αρμενία και τις άλλες τέσσερις χώρες της ε, ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πλην της Λευκορωσίας στην ε, συνέλευση της Euronest που θα δώσει πολύ περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες και στην Αρμενία και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για να προσπίσουν τις ιδέες τους και τα συμφέροντά τους μαζί μας και από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζουμε η προσοχή μας ε, να μην αποσπαστεί από τα προβλήματα στο Νότο, γιατί και στην Ανατολή και στην Ανατολική εταιρική σχέση έχουμε πολλά προβλήματα και ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με εκείνη η προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε κύριε Βιγγένιν. Ο κύριος Αρλάκη έχει το λόγο. Uh, Πρόεδρε, ε, σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να υποβάλω δύο σύντομες ερωτήσεις. Η μία έχει σχέση με τον Αγκόρνο Καραμπάχ με τη διένεξη στον Αγκόρο Καναπά και είναι πάρα πολύ απλή ερώτησή μου. Ποια είναι η θέση σας απέναντι στο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών ε, σχετικά με την επίλυση του προβλήματος του Αγκόρνο Καραμπάχ. Δεύτερον, όσον αφορά ε, τον ποινικό αντιδραστήρα Τζαμόρ, ο οποίος ε, έκλεισε όταν είχαμε το μεγάλο σεισμό στην Αρμενία και ξανά άνοιξε το 1993 και καλύπτει σημαντική ενέργεια της Αρμενίας. Η Αρμενία δέχτηκε να κλείσει αυτό το ποινικό αντιδραστήρα μετά από μεγάλη πίεση που ασκήθηκε τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ο αντιδραστήρας αυτός, ο πυρηνικός, είναι ο παλαιότερος ε, και ο λιγότερο αξιόπιστος ε, που κατασκευάστηκε σε πρώην κράτος της Σοβατικής Ένωσης. Εσείς παρακαλώ, τι έχετε να μας πείτε σχετικά με αυτό το θέμα. Ε, Ποιε είναι οι τελευταίε εξελίξει επ' αυτού. Ευχαριστούμε τον κύριο Αρλάκη. Λούνατσεκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ε, σας καλωσορίζω εκ μέρους των ε, Πρασίνων που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Υπάρχουν δύο θέματα που θα ήθελα να, να, να εξετάσω. Όπως υπάρχει και προηγουμένως το θέμα του πυρηνικού αντιδραστήρα που έχετε στη χώρα σας, τον Μετσαμόρ, ο οποίος, ε, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ένας από τους παλαιότερους που εξακολουθεί να λειτουργεί. Θα ήθελα λοιπόν και μάλιστα έχει ε, κατασκευαστεί πάνω σε σεισμογενή περιοχή και θα ήθελα να πω το εξή. Η δική σα η αρμόδια επιτροπή για θέματα πυρηνική ενέργεια είπε ότι μετά την καταστροφή στην Ιαπωνία ο αντιδραστήρα αυτό, ο Μετσαβόρ, είναι αρκετά ασφαλή, ότι σεισμό τέτοια κλίμακα είναι μάλλον απίθανο να πλήξει την αρμονία και δεν πρέπει να ανησυχούν οι Αρμένοι. Εντάξει, δεν το είπα ακριβώ έτσι. Εγώ το ερμηνεύω κάπω έτσι. Επίση, ο πρώην Γενικό Διευθυντή του Μετσαμόρ είπε ότι ε, το, αντιδραστήρα αυτό που είναι κοντά στο Γερεβάν δεν είναι τόσο σωστά καλυμμένος από ενδεχόμενο διαρροή. Θέλω λοιπόν να γνωρίζω από εσάς και νομίζω το 2007 αποφασίσατε ότι θέλετε να κατασκευάσετε και νέο αντιδραστήρα. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ. Υπάρχει το ενδεχόμενο να αναθεωρήσετε τη στάση σας και απέναντι στον Μετσαμόρ ε, όσο και απέναντι στην ε, καταστροφή μετά την καταστροφή στην Ιαπωνία. Γιατί δεν ξέρουμε, εφόσον είναι σεισμογενής η περιοχή αυτή, δεν ξέρουμε ακριβώς ε, ποια κλίμακας ε, θα μπορούσε να είναι ένα, το ενδεχόμενο σεισμού στο Γερεβάν. Επίσης, ε, έχετε εσείς κάποια προγράμματα για την πυρηνική ενέργεια για να μην χρειαστεί να κατασκευάσετε κάποιους καινούριους αντιδραστήρες. Το άλλο θέμα αφορά τον Αγκόρνο Καραμπάχ μιλήσατε και θα μου επιτρέψετε να είμαι ειλικρινής. Εσείς μιλήσατε ε, για την πολεμοχαρή ρητορική του Αζερβαϊτζάν και τον ε, υπερβολικό αμυντικό τους προπολογισμό. Δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό, αλλά διάβασα ότι και στην Αρμενία το 19% ε, του προπολογισμού σας είναι αμυντικές δαπάνες. Το 19% θα έλεγα και εγώ, το κρίνω υπερβολικό, ακραίο. Ποια είναι λοιπόν η δική σας η προσέγγιση. Εσείς επιρρύπτετε την ευθύνη για το πρόβλημα στο Αζερμπαϊτζάν. Λυπούμε που μιλάω ειλικρινά, αλλά ξέρετε ε, στην πολιτική δεν μπορεί κανείς ε, να επιλύσει οτιδήποτε αν ε, αποσύει τις ευθύνες του και ρίχνει το βάρος στην άλλη πλευρά. Εσείς λοιπόν, από τη δική σας τη σκοπιά, εσείς και η χώρα σας, τι μπορείτε να κάνετε για να άρετε το αδιέξοδο το οποίο έχει διαμορφωθεί στις σχέσεις των δύο χωρών. Παραδείγματο χάρη, θα μπορούσατε να φανταστείτε να δώσετε κι εσείς ένα δείγμα καλής θέλησης με το να αφήσετε ελεύθερες κάποιες από τις κατεχόμενες περιοχές γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχ και μετά να ακολουθήσουν οι άλλοι. Και κάτι άλλο, στην Αρμενία υπάρχει μεγάλη διαρροή εγκεφάλων. Πολλοί νέοι Αρμένοι φεύγουν γιατί αισθάνονται ότι δεν έχουν μέλλον στη χώρα τους. Και τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε για να τους κρατήσετε εκεί γιατί νομίζω ότι τους χρειάζεστε. μου. Προσθέθηκαν και άλλοι ερωτώντες. Ο χρόνος φεύγει γρήγορα. Τρία λεπτά παρακαλώ ο καθένας. Ο κύριος Κέλαμ. Uh, Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά με την έλευση σας εδώ γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε αξίες και η Αρμενία είναι η αρχαιότερη χριστιανική χώρα και εξασφαλίζει τη συνέχεια αυτών των αξιών. Ως εκ τούτου σας αξίζει μια ιδιαίτερη θέση στις σχέσεις μας. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την Αρμενία στην συνέλευση της Euronest που θα αρχίσει να συνεδριάζει όπως ανέφερε και ο κύριος Βιγκένιν. Μας αναφέρατε κάποιες μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντικές σας και θα θέλαμε τη γνώμη για το πού μπορεί να σας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές. Άλλο θέμα είναι οι επενδύσεις στην Αρμένια ποιο είναι ο φόρο εισοδήματο, ποιε είναι οι προποθέσει ε, για τι επενδύσει, τι φόρο εισοδήματο καταβάλουν οι επιχειρήσει στην Αρμενία. Σα ευχαριστούμε κύριε Κέλαμ. Ο κύριο Νταφ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε. Ποιος είναι ο πυρήνας του ιστορικού αλλά και του σύγχρονου προβλήματος με την ε, Τουρκία. Την ιστορία την ξέρουμε, αλλά δώστε μας μια επίκαιρη προοπτική αυτών των προβληματικών σχέσεων με την Τουρκία. Πιστεύετε ότι η επιρροή της αρμενικής διασποράς που είναι πραγματικά μεγάλη, γιατί η αρμενική διασπορά είναι εγκατασπαρμένη παντού στον κόσμο και έχει και μεγάλες διαστάσεις. Πιστεύετε ότι αυτό εμποδίζει τη δυνατότητα της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου σας να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία και να εξυγχρονίσουν τις ε, θέσεις τους. Γιατί μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι η θέση των απόδημων Αρμενίων της αρμενικής διασποράς είναι πολύ πιο δηλητηριώδης, ε, αντιδραστική και εθνικιστική από ότι τα μηνύματα που εκπορεύονται από τη διοίκηση της χώρας και τα μηνύματα που ακούμε εντό τη χώρα. Για τρία λεπτά, κύριο Τάνοκ. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Σα καλώ ορίζω Έχουμε ξανασυναντηθεί και δεν θέλω να πούμε αυτά που είπαμε ήδη προηγουμένως καταρχήν χαιρετίζω το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησής σας που έδειξε δυνατότητα ανάκαμψης μετά από σημαντική συρρήγνωση της οικονομίας σας το 2008 και αν η οικονομία μπορούσε να επιλέξει πού θα βρίσκεται στο ενηφίλιο, θα ήθελε να είναι κάπου αλλού αντί περιστοιχισμένη από δύσκολους γείτονες στο Ιράν, τη Σοβιετική Ένωση στην Τουρκία είσαστε ε, βασικοί και ε, για την ενεργειακή ασφάλεια και για την γεωπολιτική σταθερότητα. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε εσείς για να συνδράμετε την ε, κατάσταση. Ήμουν υπέρ της πολιτικής γυτνιάσεως και πίστευα ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την κοινωνία των πολιτών στον παρα Καραμπάχ και εφόσον ε, χρηματοδοτούσαμε την Απκασία, τη Νότιο σετία και ε, λόγω κάποιας πιέσεως ε, δεν υπήρχε αυτή η κίνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον αγώνο Βαραγκάς. Πιστεύω ότι η φιλοπόλεμη ρητορική για, από τον Μπακού που είναι πλούσιο με πετροδολάρια ε, ε, ε, έχει επηρεάσει γιατί είσαστε μια μικρή οικονομία ίσως είστε υποχρεωμένος να καλύψετε με 19% του προϋπολογισμού σας την, τις πολεμικές δαπάνες διότι δυστυχώς ως επιτοπλίστων οι επιλύσεις των διαφορών είναι στρατιωτικές και δεν μπόρεσε να υπάρξει όμως όμως στρατιωτική λύση στον αγόρνο Παραμπάχ πρέπει να υπάρξει μια ειρηνική λύση και πλέον τι κάνουν οι σύμμαχοί σας η Γαλλία κάνει επαρκείς κινήσεις μήπως η ύπατη εκπρόσωπος μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω διότι η θέση που είχε ο Πίτερ Σάμνομπι για τον Νότιο Κάφκασο και κατεργήθη θα μπορούσε να συμβάλλει Υπάρχει ένα υπερεθνικό ρόλο στην περιοχή για να επιλύσει θέματα σαν τον Αυγόνο Καραμπάθ αφού κατεργήθηκε λέγεται ότι κάποιος θα αναλάβει όλες τις διαφορές ε, και προς την Τρανιστρία και προς τη Μολδαβία και όλη την περιοχή. Μήπως λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη οικονομική ε, υλοποίηση ή στο Νότιο Κάφκασο για να έχουμε αποτελέσματα ε, διότι εάν ε, δεν βελτιωθεί η κατάσταση και επανέλθουμε σε στρατιωτικές σειράξεις και η Δύση θα φέρει από την διακοπή της ε, προμηθείας ε, ενεργείας και θα αναρωτηθούμε γιατί δεν κινηθήκαμε πιο έγκαιρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τάνοκ και το ε, λόγο έχει ο κύριος Κυρίλοφ τρία λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κοντά μας κύριε Πρωθυπουργέ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ειλικρινείς παρατηρήσεις και την ειλικρινή παρουσίαση της χώρας σας και της σύγκρουσης. Συμφωνώ μάλλον μαζί σας ότι μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, 20 περίπου χρόνια, όπου υπήρχε απόλυτο αδιέξοδο και υπάρχει αδιέξοδο στον Αγκόνο Καραμπάχ, κάτι πρέπει να γίνει. Εσείς είπατε ότι ε, πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές ε, και στις δύο πλευρές. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί ως έχει γιατί υπάρχουν θύματα και στις δύο πλευρές. Εγώ πρέπει να σας ε, πω πρόσφατα άκουσα ότι υπήρξαν και δολοφονίες ε, στο Γερβάν από ελεύθερους ε, σκοπευτές. Ε, η κατάσταση λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο. Εσείς είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο. Μέχρι τώρα μπορεί να μην τα καταφέραμε καλά, αλλά η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε κάτι να κάνουμε. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Λούνατσεκ, στην περίπτωση που συμφωνήσετε πάνω σε ένα ρηψταραλέο και επικοδομητικό βήμα. Παραδείγματο χάρη, να αποσυρθείτε από κάποιες κατεχόμενες περιοχές γύρω από τον Αγκόνο Καραμπάχ. Βεβαίως και χρειάζεστε εγγύησει, γιατί ξέρετε εγώ το συζήτησα αυτό ε, άτυπα με κάποιους ε, πολιτικούς σας. Ε, πιστεύετε ότι αν αποσυρθείτε εσείς ίσως τις περιοχές αυτές καταλάβει το Αζερμπαϊτζάν. Ερωτώ όμως, θεωρείτε ότι είναι προς το συμφέρον σας να καταφύγετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω ακόμα και στη Ρασία, να τους ζητήσετε να τοποθετήσουν εκεί δυνάμεις ειρηνευτικές για να επιτευχθεί η λύση. Πριν από μία εβδομάδα στη συνάντηση με τον Μετβέντεφ ε, διαπίστωσα τι έγινε ακριβώ εκεί γιατί διαπίστωσα ότι δεν ήταν και τόσο ήταν κατά κάποιον τρόπο αρνητικές οι παρατηρήσεις που έγιναν και από τις δύο πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προτίθεται να στηρίξει το ειρηνικό μέλλον σε αυτή την περιοχή, τις ειρηνικές εξελίξεις, γιατί ενδιαφερόμαστε όλοι για αυτό το κομμάτι της γης. Ο κύριος Σαλαφράγκα, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και να σας πω ότι καλό θα ήταν η σημερινή σας παρουσία εδώ να μην είναι και η τελευταία, αλλά να αποτελέσει την απαρχή μια σειρά επαφών που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε το διάλογό μας και να είμαστε επικοδομητικοί για να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ μας προκλήσεις. Και όταν μιλώ για την έλευση σας εδώ στην Επιτροπή, δεν μιλάω μόνο για την παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά γιατί όχι και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως έχουν κάνει και εκπρόσωποι άλλων χωρών της περιοχής. Με ενδιαφέρει κύριε Πρωθυπουργέ η γνώμη σας για το εξής. Τι θα γίνει με τις ε, επόμενες εκλογές, γιατί του χρόνου έχετε νομοθετικές εκλογές και τον επόμενο χρόνο προεδρικές εκλογές τις ε, εκλογικές και μετακλογικές ε, συγκρούσεις που είχατε στη χώρα σας, ε, σκόπι μου θα ήταν οι επόμενες εκλογές να γίνουν απρόσκοπτα, με διαφάνεια, με ομαλότητα, ώστε πραγματικά αυτό που θα προκύψει από τις κάλπες να είναι η πραγματική βούληση των Αρμένιων πολιτών. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτές τις επερχόμενες εκλογικές διαδικασίες. Κάποιος συνάδελφος μίλησε για το βάρος που έχει στη χώρα σας η γνώμη της διασποράς, η απόδημη Αρμένη πραγματικά δεν γνωρίζω τον αρμενικό εκλογικό νόμο και δεν ξέρω αν οι απόδημοι Αρμένοι έχουν δικαίωμα ψήφου, γιατί πραγματικά είναι σημαντική η αρμενική διασπορά και δεν ξέρω πώς συμμετέχει στην, ε, στις εκλογές. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε τι προσδοκείτε από την ε, Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποιο βαθμό αυτή η Συμφωνία Σύνδεσης θα μπορούσε να σας βοηθήσει όχι μόνο για να ευαθύνεται το σημαντικό θέμα που έθεξε ο κύριος Κέλλαμ που είναι το θέμα των αξιών και που φυσικά αποτελεί τη βάση όλων των συμφωνιών σύνδεσης και το θεμέλιό τους, αλλά για να σας βοηθήσει να υπερβείτε και την ε, δυσχερή οικονομική κατάσταση που από το 2008 σας ταλανίζει, όπως είπε και ο κύριος Στάνοκ. Επίσης, με ενδιαφέρουν και εξελίξεις το θέμα στη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ και οι σχέσεις σας με τη Ρωσία. Ο τελευταίος προελής ρώτησε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί καλύτερα και περισσότερο ώστε να βοηθήσει μια ειρηνική λύση, επίλυση μάλλον του, της σύγκρουσης αυτής. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα. Για τρία λεπτά ο κύριος Κούκαν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ και σας καλωσορίζω θερμά κύριε Πρωθυπουργέ. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω και τα μέλη της αντιπροσωπείας σας. Εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτά που μας είπατε, ε, το πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση στη χώρα σας σε νυφάλια και πολύ συγκεκριμένα και ρεαλιστικά αυτά που μας είπατε. Οι συνάδελφοι νομίζω ότι εξάντλησαν όλες τις ε, ερωτήσεις που θα μπορούσαν να υποβληθούν, τα προβλήματα που αφορούν στη χώρα σας. Εγώ απλά θα αναδιατυπώσω Κάποιε ερωτήσει. Δηλαδή, όταν συζητάμε την κατάσταση σε άλλε περιοχέ του κόσμου, στην Ευρώπη, τίνουμε πάντα να υπογραμμίζουμε τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης. Βεβαίως η κατάσταση ίσως στην περιοχή σα είναι λίγα και διαφορετική λόγω του ότι υπάρχει μια ανήσυχη θα τη χαρακτήριζα ε, σχέση, διμερή σχέση με άλλες χώρες και προσβλέπω στις απαντήσει σα. Ε, στις ερωτήσεις του κυρίου Νταφ όσον αφορά στη σχέση της χώρας σας με την Τουρκία λαμβανομένης υπόψης της ιστορίας που έχει προηγηθεί του παρόντος στη χώρα σας. Πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθούν οι σχέσεις με την Τουρκία. Κάτι τέτοιο ε, θα ήταν εποφελές ε, για την εξωτερική πολιτική της χώρας σας. Επίση, θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον κατά την άποψή σα είναι ρεαλιστικό να σκέπτεται κανείς ότι θα μπορούσε στην ε, περιοχή σα και στη χώρα σας να υπάρχει μια ουσιαστική περιφερειακή συνεργασία. Ευχαριστούμε και ο κύριος Βάγκολ για τρία λεπτά θα ολοκληρώσει τις ερωτήσεις. Πρόεδρε, και για μένα, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω εδώ ε, σήμερα. Ε, σας συγχαίρω για τις προσπάθειες που καταβάλει η χώρα σας ε, προς την κατεύθυνση των οικονομικών ε, μεταρρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων της δικαστικής εξουσίας. Ήμουν πρόσφατα στον Μπακού ε, και παρακολούθησα μια συνάντηση, μια συνδιάσκεψη οργανώθηκε από την Επιτροπή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είχαμε εκεί εκπροσώπους και δικών σας ΜΚΟ, οι οποίοι είχαν έτσι ένα πολύ φιλικό διάλογο με τους συναδέλφους τους από το Αζερβαϊτζάν. Έτσι λοιπόν και εγώ Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή όλες οι άλλες ερωτήσεις έκαναν ήδη στην συνάδελφοί μου. Να ρωτήσω λοιπόν, δεν πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να ε, επενδύσετε περισσότερο στο να υπάρξει ένας απευθείας διάλογος με το Αζερβαϊτζάν τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο, σε επίπεδο ε, κοινωνίας των πολιτών. Ένας διάλογος που θα μπορούσε να αλλάξει τη φύση και το μοντέλο μέσα στο οποίο εντάσσονται τα προβλήματα. Στον Πακού άκουσα πολλές αιτιάσεις εις βάρος ε, της ε, χώρας σας, ε, περίπου όπως τα είπατε και εσείς σήμερα. Άκουσα αιτιάσεις του Μπακού, του Τερμπατζάν που έχουν σχέση με την στρατιωτική απειλή από εσά. Βεβαίως οι ε, εταίροι μου ε, στον Πακού λένε, μου είπαν ότι τάσσονται ανεπιφύλακτα κατά της ε, στρατιωτικής λύσης. Θα λοιπόν να σας ερωτήσω το εξής εσείς βλέπετε να υπάρχει μια δυνατότητα για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο σε αυτό το διάλογο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η ομάδα Μίνσκ δεν αρκεί. Εδώ και 15 χρόνια ε, δεν έχει επιτύχει τίποτα το σημαντικό. Ε, χρειάζεται λοιπόν ε, φρέσκο αίμα και νέες ιδέες να πω το εξή τελειώνοντα. Έχω την εντύπωση ότι ε, σε αυτό το πολύ περίπλοκο σκηνικό που επικρατεί στην περιοχή και που περιγράψετε εσεί και οι συνάδελφοί μου, έχω την εντύπωση λοιπόν ότι εκεί οι μικρέ χώρε ε, πολύ συχνά είναι θύματα των ε, συμφερόντων των μεγαλύτερων συμμάχων και εταίρων που μερικές φορές είναι και επικίνδυνη. Ίσως λοιπόν ε, θα πρέπει να μην επαφίεστε μόνο σε μία μεγάλη χώρα που σας υπόσχεται βοήθεια αν τελικά ε, προκύψει, εξελιχθούν τα πράγματα σε πραγματική σύγκρουση. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος ε, και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο ε, στον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. հարցերի համար Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια ε, τα οποία έγιναν. Σε 12 λεπτά τώρα θα ε, αποπειραθώ να απαντήσω στα ερωτήματα που μου ετέθησαν συγκεντρώνοντας τις ερωτήσεις σε επιμέρους κεφάλαια. Σχετικά με το ορεινό Καραμπάχ. Καταρχήν διαστάνθηκα ότι θέλετε να μας βοηθήσετε στο ζήτημα του ορεινού Καραμπάχ ώστε να επιληθεί το ταχύτερο δυνατό. Και για τούτο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Και θέλετε να ακούσετε την άποψή μου για το πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να επιληθεί το ζήτημα. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσουν. Σε κάθε σύγκρουση οι δύο πλευρές έχουν διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο επίλυσης του ζητήματος. Και συνεπώς οι δύο πλευρές θα πρέπει να καθίσουν σε διαπραγματεύσεις και να καταλήξουν σε συμφωνία. Όταν όμως οι δύο πλευρές κάθονται γύρω από ένα τραπέζι αλλά σκέφτονται ότι το ζήτημα θα επιληθεί όχι γύρω από αυτό το τραπέζι, πάνω σε αυτό το τραπέζι, αλλά εκτός αυτού του χώρου, τότε δεν είναι δυνατόν να βρεθεί λύση. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ως προς την επίλυση του ορεινού Καραμπάχ. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε. Δεν υπάρχει άλλη αναλλακτική πέραν της ειρηνικής επίλυσης. Αν λοιπόν ισχύει τούτο, η δική μου απάντηση για το ποια μπορεί να είναι η ουσιαστική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απάντησή μου είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ξεκάθαρα να πει στις δύο πλευρές ότι εάν οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές αποπειραθεί να επιλύσει το ζήτημα με βία μέσα, η διεθνής κοινότητα θα επιβάλλει τα, τις αυστηρότερες κυρώσεις και αν υπάρξει από πλευράς διεθνούς κοινότητας τέτοια ξεκάθαρη δήλωση ότι δηλαδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέραν της ειρηνικής επίλυσης τότε σας διαβεβαιώνω ότι ασφαλώς οι διαπραγματεύσεις μπορούν να καταλήξουν σε επιτυχία. Αυτό το οποίο επιτέλεσε η ομάδα του Μίνς και η πρόοδος που έχει σημειωθεί και το λεπτο, έργο το οποίο ε, έχουν υλοποιήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία και Γαλλία στο πλαίσιο της ομάδας του Μίνσκ νομίζω ότι έχουν δημιουργήσει το απαραίτητο πλαίσιο ώστε να μπορέσει το ζήτημα του ορεινού Καλαμπάχ να επιληθεί με ειρηνικά μέσα διότι οι ε, συμβιβαστικές προτάσεις που έχουν γίνει μπορούν να αποτελέσουν βάση για την περαιτέρω εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Έτσι λοιπόν, αν υπάρξει από πλευράς διεθνούς κοινότητας τέτοια δήλωση ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να επιληθεί με ε, στρατιωτικά μέσα, τότε ασφαλώς και οι δύο πλευρές μπορούν να περιορίσουν τις ε, ε, στρατιωτικές δαπάνες. Αλλά στο βαθμό που η μία εκ των δύο πλευρών βλέπει ότι έχει πολλές πιθανότητες να λύσει το ζήτημα με στρατιωτικά μέσα και καταβάλει προσπάθειες και δαπανά τεράστια ποσά, τότε ασφαλώς δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία η ειρηνική επίλυση. Δεύτερον, πώς μπορεί να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα αυτό. Εάν οι δύο πλευρές έχουν διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της επίλυσης του ζητήματος ε, τούτο σημαίνει ότι έχουν διαφορετική αίσθηση ως προς το δίκαιο, ως προς την δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με ένα σύστημα αξιών. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι υπάρχει συγκεκριμένη συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως ανέφερα, είναι η ενιαία πλατφόρμα αξιών στην περιοχή μας. Αν λοιπόν συμφωνήσουμε πάνω στις θεμελιώδεις αξίες, τότε θα είναι εύκολο να επιληθούν όλα τα ζητήματα που εκκρεμούν, όλες οι σειράξεις. Και εγώ βλέπω μόνον ένα δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Τουρκία και Αρμενία έχουν δηλώσει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ζωτική σημασία η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι τέσσερες χώρες προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες μας οδηγούν προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, οι δεδηλωμένες ε, αξίες, αυτές οι οποίες δηλώνουμε ότι πιστεύουμε, διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα. Υπάρχει δηλαδή τεράστια διαφορά μεταξύ αυτών που δηλώνουμε και αυτόν που στην πράξη εφαρμόζουμε. Έτσι λοιπόν είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση ε, θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζει διαδραματίζουν οι μεταρρυθμίσεις και η εφαρμογή των ευρωπαϊκών αξιών. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη της ενίσχυσης, της αρρωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, να γίνουν οι σε βάθος μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Βεβαίως σημειώθηκε πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως σημειώθηκε πρόοδος στην ε, υλοποίηση, στην εφαρμογή αυτών των αξιών. Ε, απαιτείται όμως κάτι ακόμα περισσότερο. Αν αυτό επιτευχθεί, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να οδηγηθούμε και σε λύση. Το τρίτο ζήτημα το οποίο ανησυχεί πολλούς είναι το ζήτημα της μονάδας πυρηνικής ενέργειας, η διακοπή λειτουργίας του και η κατασκευή μιας νέας πυρηνικής μονάδας, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στην Ιαπωνία το θέμα καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρο. Διότι σε όλες τις χώρες όπου λειτουργούν μονάδες πυρηνικής ενέργειας αυτή τη στιγμή διεξάγονται ε, έντονες ε, συζητήσεις. Και εμείς εξετάζουμε το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε την ασφάλεια τη δική μας μονάδα πυρηνικής ενέργειας και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με όλους τους διεθνείς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων. Έχουμε ανοιχτή και διαφανή συνεργασία και αφενός εφαρμόζουμε ένα πολύ ξεκάθαρο και διαφανές πρόγραμμα εφαρμογής των βασικών θεμελιωδών αρχών ασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξηθεί ο βαθμός ασφάλειας. Και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την βοήθεια αυτή και Βεβαίω, όπως σε όλες τις χώρες, έτσι και εμείς στην Αρμενία, για μία ακόμα φορά εξετάζουμε με μεγάλη σοβαρότητα το ζήτημα της ασφάλειας της μονάδας του Μετζαμόρ. Το άλλο ζήτημα είναι οι σχέσεις με την Τουρκία. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι προς το συμφέρον μας να επιτύχει η Τουρκία το στόχο της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μας συμφέρει να έχουμε μια Τουρκία δημοκρατική, εξελιγμένη, ε, ε, μια γειτονική χώρα η οποία θα εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες διότι αυτό θα συμβάλλει τόσο στην ασφάλεια της περιοχής και θα συμβάλλει επίσης και στην δημιουργία πιο ευνοϊκών συνθήκων για συνεργασία με την Αρμενία. Η δική μας πολιτική τα τελευταία 20 χρόνια δεν μεταβλήθηκε, παραμένει η ίδια. Εμείς είμαστε έτοιμοι, χωρίς προϋποθέσεις, να ε, εγκαθιδρύσουμε διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία και, τουρ... σχέσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν ε, τους γείτονες. Απόδειξη τούτου είναι ότι με τρόπο τολμηρό θα έλεγα πήγαμε στην Ελβετία και υπογράψαμε τα δύο πρωτόκολλα και ο πρόεδρος της χώρας μας δήλωσε ότι είμαστε έτοιμοι να επικυρώσουμε αυτά τα δύο πρωτόκολλα. Επιπλέον το συνταγματικό δικαστήριο της ε, ε, Αρμενίας επικύρωσε, της Αρμενίας επικύρωσε και επιβεβαίωσε την απόφαση αυτή. Δυστυχώς όμως δεν ανταποκρίθηκε η Τουρκία σε αυτό. Η Τουρκία δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει σε καθιέρωση φυσιολογικών σχέσεων με την Αρμενία χωρίς προϋποθέσεις. Το επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με τις αρμενικές κοινότητες. Ο αρμενικός λαός είναι ένας ενιαίος οργανισμός και είναι σφαλμένη η εντύπωση ότι μπορεί το ένα κομμάτι, ή το ένα σκέλος ενός λαού να έρθει σε αντιπαράθεση με το άλλο σκέλος αυτού του λαού. Αυτό είναι εντελώς αφύσικο. Στον κόσμο υπάρχουν πολλοί λαοί που διαθέτουν διασπορά. Και αν οι εκπρόσωποι αυτής της διασποράς ταυτίζονται ή ε, εμφανίζονται ως ε, τέκνα ε, ενός ενιαίου λαού, αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά τους. Βεβαίως τούτο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ε, ποικιλομορφία απόψεων στους κόλπους του αρμενικού λαού. Και τούτο ισχύει και εντός της Αρμενίας και εκτός Αρμενίας στη διασπορά. Για το πώς δηλαδή μπορούν να διευθετηθούν οι αρμενοτουρκικές σχέσεις και εντός της Αρμενίας υπάρχει αντιπολίτευση και εμείς απολέσαμε ε, ένα από τα κόμματα της ε, ε, κυβερνητικής συμμαχίας ακριβώς επειδή διαφωνούσε με την υπογραφή των πρωτοκόλων και να, υποβάλουμε τα πρωτόκολλα σε επικύρωση από το κοινοβούλιο μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η διασπορά είναι κατά, ενώ η Αρμενία είναι υπέρ. Εντός ε, του αρμενικού λαού, στους κόρπους του αρμενικού λαού υπάρχουν διαφορές απόψεων. Το άλλο θέμα είναι οι σχέσεις μας με τον στρατηγικό μας εταίρο που είναι η Ρωσία. Η Ρωσία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην δημοκρατία της Αρμενίας. Και επιπλέον να πω ότι υπάρχουν εγκατεστημένες ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και τούτο είναι ε, συνειδητή και σταθμισμένη επιλογή της ε, κυβέρνησης της Αρμενίας. Διότι στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλές μη διευθετημένες πολλά μη διευθετημένα μη ε, ε, ζητήματα, ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί, εμείς έχουμε ανάγκη να διασφαλίσουμε την φυσική ασφάλεια του λαού μας. Την ασφάλεια του λαού μας. Ε, την ασφάλεια ενός λαού που έχει γνωρίσει γενοκτονία και που στο υποσυνείδητό του το ζήτημα της ασφάλειας έχει θεμελιώδη, ουσιαστική σημασία. Όταν λοιπόν ε, ε μάλλον πότε ε, θα χρειαστεί να ή θα είναι δυνατόν να αποσυρθούν αυτές οι δυνάμεις ε, από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Όταν πλέον δεν θα υπάρχει ανάγκη παρουσίας τους, δηλαδή μέσω των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Ε, εάν υπάρξει επιτυχία, εάν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών, τότε δεν θα υπάρχει ανάγκη και παρουσίας των στρατιωτικών δυνάμεων. Έρχομαι τώρα στο θέμα των δασμών και των φόρων. Ε, Ρωσία, Καζακστάν και Λευκορωσία όπως ελέγχθη, ήδη συζητούν και το, και το θέμα συζητείται και στην κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών και το ζήτημα έχει συζητηθεί και με την Αρμενία. Η δική μας θέση είναι η εξή. Η Αρμενία πρόκειται να γίνει μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Εμείς δηλαδή έχουμε συμπεριλάβει και εφαρμόζουμε όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την ένταξή μας στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Το ίδιο επιδιώκει και η Ρωσία και προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλει ουσιαστικές και σοβαλές προσπάθειες. Στη διεθνή πρακτική δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα όπου οποιαδήποτε χώρα ε, οποιαδήποτε χώρα που δεν έχει ε, σχέσεις με τις ε, γειτονικές χώρες και δεν έχει ρυθμίσεις δασμολογικές με τις χώρες αυτές να ενταχθεί στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Τούτο σημαίνει ότι η Τελωνιακή Ένωση, ε, στην Τελωνιακή Ένωση ε, Ρωσίας, Καζακστάν ε, και Λευκορωσίας η Αρμενία δεν μπορεί να ενταχθεί αν δεν ενταχθεί η Γεωργία. Ωστόσο το σενάριο σήμερα είναι το εξής. Εμείς επιδιώκουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και γι' αυτό ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε μάλλον θα καταστούμε μέλη, μέλη ε, αυτή τη ευρεία και συνεκτική ζώνη ελευθέρου εμπορίου και προς αυτή την κατεύθυνση κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Έρχομαι τώρα στο θέμα τη ε, Euronest. Η δική μας θέση είναι η εξή. Εμείς συμμετείχαμε και θα συμμετάσχουμε στη διαδικασία αυτή, διότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία αυτή, διότι βλέπουμε ότι διαμορφώνεται μια πολύ σημαντική πολιτική πλατφόρμα όπου οι βουλευτές θα μπορούν να εξετάζουν θέματα τα οποία απασχολούν αλλήλους και τούτο μπορεί να συμβάλλει ε, προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης. Εμείς λοιπόν ε, είμαστε υπέρ της δημιουργίας αυτού του οργάνου. Ε, στη δημοκρατία της Αρμανίας βεβαίως υπάρχουν ακόμα εκκρεμή ζητήματα. Και ένα βασικό θέμα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι το εξής. Ε, δεδομένου ότι έγιναν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις εκλογές. Σε ένα χρόνο έχουμε κοινοβουλευτικές εκλογές και εμείς πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι εκλογές αυτές να διεξαχθούν ε, με βάση τις αποδεκτές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Κατά τη γνώμη μου η καλύτερη απάντηση στα ερωτήματα αυτά θα είναι η εξής. Θα πρέπει εμείς να δώσουμε νέα όθηση στο πακέτο ή στο σχέδιο μεταρρυθμίσεων που υλοποιούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να καταστούμε μια χώρα η οποία λειτουργεί ε, δημοκρατικά, ελεύθερα και σύμφωνα με τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Όσο πιο γρήγορα ε, υλοποιηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις τόσο γοργότερα θα αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνησή μας και τούτο θα αποτελέσει και την εγγύηση, εγγύηση για τη διεξαγωγή πιο διαφανών, ε, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών το 2013. Δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ εξάντλησα το χρόνο που μου είχε διατεθεί Και θα ήθελα για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που επιδείξατε, τις απόψεις που διατυπώσατε και τα ερωτήματα που θέσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ γιατί νομίζω ότι η αντιδράση των συναδέλφων ήταν πολύ θετική και η παρουσία σας χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ειλικρίνεια και πολλές πλήρεις πληροφορίες. Θέλουμε να σας, ευχαριστούμε, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία εις την συνέχιση της εργασίας σας, ιδίως κατά την επίσκεψη στο Κοινοβούλιο για να μας υποκινήσετε να εμπλακούμε περισσότερο περισσότερο στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα άλλα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν εδώ. Ελπίζουμε ότι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε θα υπάρχει ένα άλλο θετικό βήμα προς τα εμπρός. Σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Για πέντε λεπτά θα διακοπεί η συνεδρίαση προτού φτάσει ο Επίτροπος Φίλε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ λάβατε θέσεις γιατί πρέπει να συνεχίσουμε. Κύριε Επίτροπε, όπως ε, ήθιστε, εσείς ε, είσαστε πάντα ε, παρόν στις σημαντικές στιγμές της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής λόγω των αρμοδιοτήτων που έχετε αναλάβει και έχουμε διαπιστώσει ότι σέβεστε ιδιαίτερα τη δική μας τη δουλειά. Ας ε, συνεχίσουμε λοιπόν από εκεί που είχαμε σταματήσει πρόσφατα. Σήμερα θα μας παρουσιάσετε την κοινή ανακοίνωση ε, που έλαβε χώρα με τον ε, άλλο αντιπρόεδρο, τον Αρμόδιο, σχετικά με την ε, συνεργασία στο Νότο, την ανακοίνωση που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η δική μας λοιπόν Επιτροπή, όπως όλοι γνωρίζουν, παρακολουθούν την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στράτευση. Σήμερα το πρωί εγκρίναμε δύο ψηφίσματα, το ένα αφορά στην διάσταση του Νότου και το άλλο στη διάσταση προς Ανατολάς, ανατολική εταιρική σχέση. Ε, αυτές λοιπόν, αυτά τα δύο ψηφίσματα υπογραμμίζουν τη σημασία ε, που έχουν οι δικέ μας οι εξωτερικές ε, σχέσεις. Και επίσης αναφέρουν και πιο συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν σχέση με ε, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το προχωρισμένο αυτό καταστατικό ή ο κανονισμός. Θα έχετε φαντάζομαι ενημερωθεί ότι η δική μας Επιτροπή αποφάσισε να συστήσει μια ομάδα ελέγχου που αφορά στην κατάσταση ε, στη Νότια Μεσόγειο. Και με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε να ε, εξοικειωθούμε, να αξιολογήσουμε τη σημασία των πράξεων που αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα τις ε, τελευταίες εβδομάδες ε, στην περιοχή αυτή. Μιλάμε για μια ε, κατάσταση δημοκρατικής μετάβασης, μετάβαση δημοκρατικής, εκδημοκρατισμό. Όπως πάντα λοιπόν περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς απόψεις που θα είναι πολύ χρήσιμες για τη δουλειά μας. Ίσως μπορείτε να παραμείνετε στα 10-15 λεπτά. Αν το κάνετε αυτό θα σας είμαι πραγματικά ευγνώμων κύριε Επίτροπε. Έχετε το λόγο. Άντε, καλύτερα προς το 15, όχι προς τα 10 λεπτά. Μπορείτε να έχετε χρόνο. Thank you very much. Uh, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και φυσικά ανυπομονώ για την ε, ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα παρακολούθησης για την Νότια Μεσόγειο που αναφέρατε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, είχα έρθει εδώ τελευταία φορά στις 28 Φεβρουαρίου και τότε, από τότε είχαμε πει ότι τα συμβάντα στην Βόρεια Αφρική έχουν ιστορικές διαστάσεις. Και είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδοκιμάσει και να καλωσορίσει αυτές τις αλλαγές και την ελπίδα τους για καλύτερη ζωή στην περιοχή με περισσότερο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πλουραλισμό, κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και τις θεμελιώδεις ελευκαιρίες που βρίσκονται στον πυρήνα των δικών μας αξιών. Είπα πρόσφατα ότι τα πρόσφατα γεγονότα έδειχναν ότι οι επιθετικές ε, ε, δηλώσεις δείχνουν ότι μια χώρα δεν είναι έτοιμη για δημοκρατία. Και ένα άλλο επιχείρημα που ακούσαμε είναι ότι η δημοκρατία είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Αυτό αληθεύει. Και... Αλλά οι βαθιές δημοκρατικές αλλαγές που ζητάει ο λαός της περιοχή, στην περιοχή δεν γίνονται εν μία νυχτή. Γνωρίζουμε ότι ο εκδημοκρατισμό είναι μια εξελικτική διαδικασία και ένα συνεχής αγώνας Αυτό όμως δεν θα πρέπει να γίνει άλοθη η δικαιολογία για την επιβράδυση των μεταρρυθμίσεων. Και το μήνυμα τη περιοχή είναι σαφέ. Ήγηκε η ώρα για να αρχίσει το έργο της μεταρρύθμισης και από τη στιγμή που ξεκίνησε θα πρέπει να επιταχυνθεί. Και στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή και είπατε Εκπρόσωπος ε, υιοθέτησαν μια κοινή ανακοίνωση που θεσπίζει κάποια σχέδια για την αναθεώρηση της συνεργασίας μας με χώρες της Νοτιού Μεσογείου προκειμένου να δημιουργήσουμε μια νέα εταιρική σχέση που θα στηρίζει τις αλλαγές. Η ανακοίνωση προβλέπει κάποια βήματα, φέρετε τα βήματα που έγιναν μέχρι τώρα και τα, τους μηχανισμούς που έχουμε για να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις, ε, υποστηρίζοντας ε, τη μετάβαση στην Τινησία και την αποτροπή της ανθρωπιστικής κρίσης ε, στη, Λιβύη. στη Λιβύη. Συγγνώμη. Επίσης η ανακοίνωση προβλέπει το πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια νέα εταιρική σχέση που θα στηρίζεται σε μια προσέγγιση που θα δίνει ενάυσματα και θα βοηθά οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της χώρας της περιοχής. Θα προωθήσουμε τώρα τη συνεργασία σε τρεις κατευθύνσεις. Θα υποστηρίξουμε φυσικά τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τη δημιουργία θεσμών. Θα προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε την κοινωνία των πολιτών και να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα και θα προωθήσουμε μια οικονομική ανάπτυξη που θα είναι συμμετοχική και δεν θα αποκλεί κανέναν. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα για ένα ποιοτικό άλμα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταίρων της Νοτιού Μεσογείου που ξεκινούν μια μετάβαση προς τον δημοκρατισμό. Η νέα προσέγγιση θα στηρίζεται ανεπιφύλακτα σε μια κοινή προσήλωση προς τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εταιρική σχέση για δημοκρατία και κοινή ευημερία μπορεί να στηρίζεται μόνο σε τέτοιου είδους ε, κοινέ δεσμεύσεις. Σκοπεύουμε να αναλάβουμε δράσεις προκειμένου να υποστηρίξουμε μια ανθούσα κοινωνία των πολιτών που θα συμβάλλει στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη δημιουργία δημοκρατικών δεσμών και χρηστής διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα τομέα όπου θα προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε την ενίσχυση των χωρών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διαμορφωθεί μια πλατφόρμα κοινωνίας των πολιτών, πολιτικών κομμάτων, συνδικάτων και διαφόρων ενώσεων και σωματείων. Τρει είναι οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής μας. Θέλουμε να βελτιώσουμε καταρχήν την κινητικότητα. Πρόκειται για ένα αίτημα των εταίρων μα που βρίσκεται στην καρδιά της ε, επιθυμίας μας να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή σχέσεων με αυτούς. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς ε, κινητικότητας ε, για τις ε, ανταλλαγέ μεταξύ φοιτητών, για το ελεύθερο εμπόριο και, εμπόριο και ελεύθερες υπηρεσίες, ακαδημαϊκές επαφές, επαφές κοινωνίας των πολιτών, θέματα κατάρτισης και το καθεξής. Δεύτερον, να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά. Έχουμε μια αγορά 200 εκατομμυρίων νέων καταναλωτών στη Βόρεια Αφρική με τεράστιο δυναμικό επενδύσεων, εξαγωγών και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό το δυναμικό βέβαια θα αξιοποιηθεί αν αφήσουμε τις χώρες αυτές να εξαγάγουν τα προϊόντα τους, αυτά που παράγουν. Κάτι που δεν αναφέρεται ρητά στην ανακοίνωση, αλλά αναφέρθηκε στο έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής της 11 Μαρτίου. Θα επανέλθουμε βέβαια στο θέμα αυτό, είναι θέτο χρόνο να επανεστιάσουμε τη χρηματοδότηση. Η ανακοίνωση προβλέπει μια σταδιακή προσέγγιση που θα εστιάζει την ενίσχυσή μας ενός ε, της ΕΜΠΑ, της πολιτικής γειτνίασης, αλλά και στα κεφάλαια και τη... το κεφάλαιο 4 και μετά θα δούμε και τα αποθεματικά και το μέσο ευελιξίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήδη προσπαθούν να εξασφαλίσουν την, ε, τη δανειοδότηση της ε, ΕΤΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη Νότια Μεσόγειο και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πλήρη εικόνα των αναγκών των εταίρων μας. Η ανακοίνωση βέβαια ξεπερνά αυτές τις τρεις κατευθύνσεις πολιτικής, είναι ευρύτερη. Όπως είπα και την περασμένη φορά, όταν εξετάσαμε αυτή την πρωτοβουλία, ο πρόεδρος Μπαρόζο ζήτησε από κάθε επίτροπο να εξετάσει τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με ιδιαίτερη υπερηφάνεια θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η ανακοίνωση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας των Επιτρόπων. Μάλιστα προτείνει 25 συγκεκριμένα μέτρα και απτές πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε στο έργο μας στην περιοχή της Νοτιού Μεσογείου, καλύπτοντας ένα φάσμα τομέων όπως ε, κοινωνικός διάλογος, αγροτική ανάπτυξη, μακροοικονομική υποστήριξη, ναυτιλιακή πολιτική, ευρωμεσογειακή πολιτική αεροπορία και δημιουργία μιας ε, ενεργειακής κοινότητας της Νοτιού Μεσογείου. Επίσης, ζητήσαμε από το Συμβούλιο να είναι τολμηρό υιοθετώντα δύο προτάσει που βρίσκονται επιτάπητο εδώ και καιρό. Η πρώτη αφορά την μεταρρύθμιση του κανονισμού ΕΜΠΑ, προκειμένου να αναχρησιμοποιηθούν κονδύλια περασμένων ετών, αυτά που αποκαλούμε reflows, στο μηχανισμό μας για την ευρωμεσογειακή επένδυση και την εταιρική σχέση που χρειάζεται ε, αρρωγή στις επενδύσεις και στην καινοτομία. Επίσης, ε, ζητήσαμε νέους ε, κανόνες προέλευσης ε, με τους εταίρους μας ε, της Νοτιού Μεσογείου. Μεταξύ των 25 μέτρων και πρωτοβουλειών περιλαμβάνονται και κάποιες πρωτοβουλίες που αφορούν την εξωτερική, εξωτερική μας πολιτική και το μέσο αρρωγής. Για παράδειγμα, επανεστίαση των προγραμμάτων 2011-2013 για την περιοχή και η θέσπιση ενός μηχανισμού ε, για την κοινωνία των πολιτών. Δεν ε, αφήσαμε ούτε πέτρα όρθια, εξετάσαμε όλες τις δυνατότητες και θέλουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα μέτρα. Και το Κοινοβούλιο και τα κρατημέλη, μεμονωμένα αλλά και από κοινού, θα μας βοηθήσουν στην ε, βοήθεια της υποστήριξης των πολιτικών κομμάτων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πλουραλισμού στις χώρες αυτές. Χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας για να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη αλλά και στις κυβερνήσεις στις 27 χώρες μέλη γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα μέτρα και γιατί και με ποιο τρόπο τα μέτρα αυτά θα σημάνουν ε, μια ποιοτική διαφορά στις νέες σχέσεις που θα έχουμε με τους εταίρους μας της περιοχής. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ισία και την Αίγυπτο, αλλά και σε όλη την περιοχή, συνεχίζονται με το δικό τους ρυθμό και με το δικό τους τρόπο. Κάποιες ε, ετοιμοπαράδοτες λύσεις ε, δεν λειτουργούν για όλους, ούτε θα πρέπει να τις επιβάλλουμε. Πρόκειται για διαδικασίες και μεταρρυθμίσεις που εκπορεύονται από τον ίδιο το λαό. Κάθε χώρα είναι διαφορετική και κάθε χώρα θα λάβει ε, ξεχωριστή και διαφοροποιημένη προσοχή Επίσης θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε σημαντικούς πόρους και οικονομικούς και τεχνικούς και να είμαστε έτοιμοι να διδαχθούμε από τη δική μας εμπειρία μεταβάσεων και μεταρρυθμίσεων προκειμένου να χειριστούμε αυτή τη διαφοροποιημένη μας προσέγγιση προς τις ε, χώρες της Νοτιού Μεσογείου. Αναμένεται και νέα ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και της αναθεώρησης, ε, της επανεξέτασης που είχαμε της πολιτικής αυτής το τελευταίο έτος. Οι προτάσεις μας ε, της ανακοίνωσης θα απευθύνονται φυσικά προς όλες ε, τις γειτονικές μας χώρες με ισορροπημένο τρόπο και προς Ανατολάς δηλαδή και προς τον Νότο. Θα συνεχίσουμε να δίδουμε ισορροπημένη προσοχή προς όλες τις χώρες της πολιτικής γειτονίας και θα εξασφαλίσουμε διαφοροποιημένες σχέσεις με τις εταίρους με τον τρόπο που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όχι με γεωγραφική βάση, αλλά με βάση την δέσμευση του κάθε εταίρου, την προσήλωσή του και το επίπεδο φιλοδοξίας του σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των μεταρρυθμίσεων. Θα ήθελα επ' ευκαιρία να αναφέρω ότι προβλέψαμε περισσότερο χρόνο για την ε, οριστικοποίηση της ανακοίνωσης για την πολιτική γειτονία, γιατί θέλουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά την έμπρακτη εφαρμογή της διαφοροποίησης ε, σε όλες τις γειτονικές χώρες και το πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει περισσότερα για να λάβει και περισσότερα και πώς οι δεσμεύσεις που αναλύθηκαν στην ανακοίνωση της τελευταίας εβδομάδας πώς θα εφαρμοστούν και στην πράξη. Βέβαια υπάρχουν και πολλά σημαντικά διδάγματα που θα πρέπει να αντλήσουμε από τα πρόσφατα γεγονότα σε ό,τι αφορά τις, χώρες, τις σχέσεις μας με τις χώρες ανατολικής γειτονίας. Η σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί το Μάιο. Αρχική ημερομηνία ήταν 20 Απριλίου. Έτσι θα έχουμε περισσότερο χρόνο και θα έχει χρόνο και το Κοινοβούλιο να αναλύσει τα πρόσφατα γεγονότα και μάλιστα να συνεχίσει αυτή την ανάλυση για το πώς θα επηρεάσει αυτή η ανάλυση της σχέσης μας με όλες τις ε, γειτονικέ μας χώρες. Θα ήθελα πριν ολοκληρώσω να πω λίγα λόγια για τη Μεσόγειο και για τις ε, μεμονωμένες χώρες της Νοτιού Μεσογείου. Γιατί την Ισία, η μεταβατική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει κάποια θετικά βήματα, τα πολιτικά κόμματα έχουν, ε, είναι πια νόμιμα και η ελευθερία του συνεταιρίζεστε έχει γενικευθεί. Θα δημιουργηθούν με τις εκλογές νέα, θα δημιουργηθεί νέο κοινοβούλιο και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε υποστήριξη για τις δημοκρατικές αλλαγές και τη μετάβαση καθώς και αρρωγή στην προετοιμασία των εκλογών. Θέλουμε να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών και το κράτο δικαίου. Θέλουμε να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε και την τινησιακή οικονομία. Στην Αίγυπτο έχουμε μόνιμες, είχαμε μόνιμες επαφές με τη μεταβατική κυβέρνηση και μάλιστα είπα ότι εκπρόσωπος κάθε Άστον θα σας ενημερώσει αργότερα για την επίσκεψη που είχε αυτή τη βδομάδα στο Κάιρο όπου μεταξύ άλλων είχε την ευκαιρία να συναντήσει και τον νέο Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών. Ευελπιστούμε ότι με τις αλλαγές αυτές θα γίνει ένα επιπλέον βήμα για μια κυβέρνηση συμμετοχική, αντιπροσωπευτική, ευρείας βάσεως και εκδηλώσαμε την προθυμία μας να αφιερώσουμε κάποιου πόρου για να υποστηρίξουμε τη δημοκρατική μετάβαση στην Αίγυπτο. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κάποιε λύσει, να απαγορεύσουμε οτιδήποτε, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε την Αίγυπτο όποτε θα είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, εντατικοποιούμε και την υποστήριξή μα προ την Αιγυπτιακή κοινωνία των πολιτών. Σε άλλε χώρε περιοχή ε, ε, διαπιστώθηκαν ε, θετικέ εξελίξει. Μάλιστα, ο βασιλιά του Μαρόκου ενήγγειλε κάποιε συνταγματικέ θεωρήσει και μεταρρυθμίσει και ένα δημοψήφισμα. Εντατικέ μεταρρυθμίσει αναγγέλθηκαν και από τον βασιλέα της Ιορδανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα προσβλέπει στην εφαρμογή αυτών των ε, εξαγγελιών προκειμένου να επιταχυνθούν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και στις δύο χώρες. Και έρχομαι τώρα στη Λιβύη. Παρά τις προφανείς διαφορές μας, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο λαός της Λιβύης αξίζει τις ίδιες ευκαιρίες για να διαμορφώσει το μέλλον του όπως έκαναν και οι γειτονικέ χώρες, οι γειτονικοί λαοί της Τινησίας και της Αιγύπτου. Στις 11 Μαρτίου το έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής υιοθέτησε μια σαφή θέση σε ό,τι αφορά τη Λιβύη και τον ηγέτη της. Θα παραμείνουμε συνεπείς με αυτή την πολιτική γραμμή και επιδιώκουμε στενό συντονισμό με τους βασικούς συνομιλητές μας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών αλλά και με τον Αραβικό Σύνδεσμο και την Αφρικανική Ένωση. Ήδη έχουμε ξεκινήσει επαφές προκειμένου να δοθεί κάποια συνέχεια στην πρόταση του, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να γίνει μια κοινή διάσκεψη κορυφής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αραβικού Συνδέσμου και Αφρικανικής Ένωσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δίνει μάχη και στο ανθρωπιστικό μέτωπο έχουμε παρουσία στα σύνορα της Λιβύης και μέχρι στιγμής έχουμε κινητοποιήσει 79 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα σκεφτόμαστε να απελευθερώσουμε και άλλα κονδύλια για ανθρωπιστική ενίσχυση. 71 εκατομμύρια ευρώ και θα συνεχιστούν και από άλλα. Ε, παρά τις εντυπωσιακέ προσπάθειες που έγιναν ήδη, η δυνατότητα εκένωσης ε, δυστυχώς υστερεί σε σχέση με την μεταναστευτική ροή και αυτό ίσως επιδεινωθεί τις επόμενες μέρες. Η κατάσταση δυστυχώς στρατητική εξελίσσεται υπέρ του Κατάφη και αυτό το παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία. Βέβαια, αναμένεται η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αδρανεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι ο συνταγματάρχης ε, Καντάφη πρέπει να φύγει και νομίζω ότι αυτό θα έχει σημαντικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την πολιτική μας απέναντι στη Λιβύη. Ενώ είναι σημαντικό να κρατήσουμε ανοιχτές τις διάβλους επικοινωνίας, θα πρέπει ταυτόχρονα να ασκήσουμε περισσότερη πίεση στο καθεστώς Καντάφη και να εξετάσουμε τις εναλλακτικέ λύσεις για τους επόμενους μήνες. Το Συμβούλιο εξετάζει τη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων εις βάρος του καθεστώτος ε, του Καντάφη, προκειμένου να μειωθούν οι πόροι που έχει το καθεστώς. Βέβαια, κάτι τέτοιο θα έχει αρνητικές συνέπειες για ορισμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς με τη θέση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιπλέον θα πρέπει να συνεχίσουμε τον εντατικό μας διάλογο με την Λιβυική Αντιπολίτευση. Και εξετάζουμε και κάποιες εναλλακτικές λύσεις και πιθανές επιχειρήσεις της ΚΕΠΑ και ΕΠΑ, συγγνώμη, της πολιτικής άμυνας, αλλά δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες εδώ. Είναι ιστορικές οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν τεράστια ευθύνη να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές και είμαι βέβαιο ότι μπορώ να υπολογίζω στη δική σα συνεργασία ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει τις κατάλληλε πολιτικές και να ενισχύσει τα υπάρχοντα θεσμικά μέσα και μηχανισμούς ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. 14 έχουν ζητήσει το λόγο. Μισή ώρα έχουμε στη διάθεσή μας ε, και θα πρέπει να απαντήσει και ο Επίτροπος. Άρα δηλαδή ε, θα πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο. Θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Φανσέρη, ο οποίος είναι αρμόδιος πρόεδρος της ε, Επιτροπής για τις σχέσεις με τις χώρες Μαγκρέπ. Θα μιλήσει για δύο λεπτά. Θέλω και λιγότερο, λέει ο ερωτών. Θα μιλήσω ακόμα λιγότερο. Κοιτάξτε, αν είχαμε ένα Όσκαρ, βραβείο Όσκαρ, ο Επίτροπος ε, θα ήταν ο πρώτος υποψήφιος εκ μέρους της Επιτροπής. Ε, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγε ώρε συζητήσαμε τα θέματα που συζητάμε εδώ και στην Ολομέλεια. Το θέμα είναι το εξή. Έχω την εντύπωση ότι εκείνα τα οποία αποφασίζουμε ισχύουν μόνο για την Τινησία διότι η Τινησία εξελίσσεται με ικανοποιητικό τρόπο ε, προς την κατεύθυνση της μετάβασης. Ε, αμφιβάλλω για την Αίγυπτο, ε, διότι το δημοψήφισμα που θα διοργανωθεί ίσως και να είναι και απλά μια αρνητική στάση απέναντι στα ερωτήματα που θα διαθούν. Για τη Λιβύη καταστροφή, πλήρης σύγχυση, αδυναμία και τίθεται σε κίνδυνο ο ρόλος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα το θέμα δεν είναι μόνο ότι θα χάσουμε την αξιοπιστία μας, αλλά και το γεγονός ότι δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε την ε, άποψη ενός ε, Καντάφη, ο οποίος ανακτά ε, τις ε, δυνάμεις του και αυτό θα είναι σημείο αναφοράς για πολλές άλλες χώρες, για την Αλγερία και τη Συρία πρέπει να τους χάνει. Δύο χώρες οι οποίες εντωμεταξύ ε, ψήφισαν κατά της no-fly zone στην Βορειοαφρική και αυτές τώρα βλέπουμε ότι στρέφονται υπέρ του Καντάφη. Θέλω λοιπόν να κάνω δύο απλές παρατηρήσεις. Υπάρχουν πράγματι κίνδυνοι. Ο πρώτος είναι να απογοητεύσουμε τις κοινωνίες πολιτών της Βορείου και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να επικρατήσει απογοήτευση ακόμα και στην κοινή γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα δει και η κοινή γνώμη ότι οι ε, κουβέντες και τα λόγια δεν έχουν καμία σχέση με τις ε, πράξεις. Και οι πρωτοβουλίες προς τον Νότο και προς τη Μεσόγειο, αυτά που είπατε, παρότι είναι σημαντικά, τίνουν, κινδυνεύουν να χάσουν όμως το πολιτικό τους βάρος. Ακόμα και η ιδέα που γνωρίζω ότι συζητείται ε, στους κόλπους της Κομισιόν κάποιας ε, αιρεσιμότητας, ευφύους αιρεσιμότητας και εκεί δεν θα υπάρχουν ε, οι συνομιλητές για να εφαρμόσουμε αυτή την αιρεσιμότητα. Ο συνάδελφος κ. Σαλαφρά. Eh, ε, ευχαριστώ και ευχαριστούμε τον Επίτροπο που είναι πάντα πρόθυμος να έρχεται στην Επιτροπή. Μας ενημέρωσε για την πρόσφατη ανακοίνωση που πολύ σωστά κάνει διάκριση μεταξύ το, της βραχυπρόθεσμης πτυχής και της μέσο και μακροπρόθεσμης πτυχής. Προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη των πολιτικών μας στην περιοχή και μάλιστα υποβάλλουμε την ανακοίνωση αυτή πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες όπως είναι αυτό το μέσο για την κοινωνία των πολιτών στην πολιτική γειτονία, το θέμα της ε, κινητοποίησης ε, για την αύξηση της κινητικότητας, ε, το θέμα των δραστηριοτήτων της ε, Τράπεζας Ανασυγκρότησης ε, και Συνεργασίας αλλά και της, τη χρηματοοικονομική στήριξη από την ΕΤΕ. Προσπαθούμε να προβούμε σε μια σταδιακή απελευθέρωση των ανταλλαγών στα πλαίσια και της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών που θέλουμε και νομίζω ότι πολύ σωστά μιλήσατε για τη δημοκρατία, για την τη συνεργασία για τη δημοκρατία και την ανάπτυξη, που είναι more for more, περισσότερο για περισσότερο, δηλαδή περισσότερη ανάμειξη αλλά και περισσότερε πολιτικέ και συνεργασία. Θα ήθελα να σα υποβάλω δύο ερωτήσει. Είπατε ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη χρηματοδότηση. Ερωτώ λοιπόν, μιλήσατε για την ενεργοποίηση του στρατηγικού αποθεματικού. Ποιε είναι οι διαστάσει, οι τάξει μεγέθου για τι οποίε μιλάμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα θεσμικό πολιτικό όργανο, δεν είναι ένα σύνολο απάτριδων γραφειοκρατών. Ε, δύο ε, κράτη-μέλη μαζί με το, με Λίβανο έχουμε, έχουν πρόταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τι αμφιβολίες υπάρχουν. Ο γιος του Καντάφη ε, ήδη καυχήθηκε ότι μέσα σε δύο μέρες ε, θα τελειώσει η κατάσταση γιατί θα καταλάβουν και, τους, ε, και τη Βεγγάζη που ήταν το προπύργιο των, της αντιπολίτευσης. Τι, ποια είναι η αντίδραση και τα σχόλιά σας για αυτές τις παρατηρήσεις. Η κυρία Ντεκαϊζέρ που αντικαθιστά τον κύριο Βιγκένινγκ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όπως και οι συνάδελφοί μου χαίρομαι ιδιαίτερος για αυτή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι να ακούω ότι, και να διαπιστώνω ότι η δημοκρατία είναι η προσμονή όλων των λαών και η κοινωνία των πολιτών ε, είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό και χρειαζόμαστε περισσότερη οικονομική δημοκρατία, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Βέβαια, ε, ο συνάδελφος Αλαφράγκα ανέφερε σημαντικές και ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει επανάσταση. Η δημοκρατία, η κοινωνία των πολιτών και η αποκλειστική κοινωνία ήταν θέματα ε, που αποτελούσαν μέρος των συμφωνιών τις οποίες είχαμε και εξυπακούοντο. Ήταν η εικόνα αυτή καθεαυτή της Ευρώπης στις σχέσεις της με τον κόσμο. Εκεί που δεν τα πήγαμε καλά είναι το να ε, υλοποιήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Μας προτείνεται λοιπόν νέες πρωτοβουλίες, να ενισχύσουμε ορισμένους στόχους, αλλά ουσιαστικά όχι. Ουσιαστικά μας προτείνεται να διορθώσουμε τα λάθη μας ποιος έκανε τα λάθη και ε, πώς. Αυτό με ενδιαφέρει εδώ διότι σε αυτήν την ανακοίνωση και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί και χαίρομαι γι' αυτό δεν κατακρίνω υπάρχει ένας μηχανισμός να ελέγξουμε τα λάθη τα οποία κάνουμε διότι πολύ μιλάμε και λίγα κάνουμε έχουμε μια πραγματική ε, γνώση των αποτελεσμάτων ξέρουμε ε, πόσο ενεπλάκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επίτευξη συγκεκριμένων συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων διότι πόσες φορές έχουμε κάνει ψηφίσματα για την Τινησία και την κυβέρνησή της πόσες φορές ε, υποδείξαμε ορισμένες καταστάσεις χωρίς να αλλάξουν θα έλεγα λοιπόν να υπάρξουν νέοι μηχανισμοί ελέγχου της ε, συνεκτικότητας των πολιτικών μας ε, των συζητήσεων που έχουμε και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε πολλά λάθη. γιατί η Λιβύη δεν θα επεκταθώ, αλλά ντρέπουμε που είμαι Ευρωπαία απόψε. Ευχαριστώ κύριος Βάγκελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι μέλος της ομάδος παρακολούθησης για την Νότιο Μεσόγειο και σήμερα συνδυάσαμε για πρώτη φορά και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε περισσότερες συναντήσεις χάρη δε στην καλή σας θέληση η οποία αποδεικνύεται από τη θέλησή σας να έρθετε εδώ και να ανταλλάξετε απόψεις με το Κοινοβούλιο θα προχωρήσουμε. Νομίζω όμως ότι η ομιλία σας ήταν ένα ρέκβιεν, ένας επικίδιος για την επανάσταση της Λιβύης για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι διακινδύνευσαν τα πάντα υπέρ της αλλαγής στη Λιβύη. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Διότι σήμερα ακούσαμε πολλές εκκλήσεις στο χώρο αυτό. Να μην εγκαταλείψουμε τους Λιβύους όπως η Ευρώπη εγκατέλειψε τους Ούγγρους το 1956, όπως εγκατέλειψε τους Ισπανούς επαναστάτες στη δεκαετία του 30. Δεν υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι η ιδέα μιας ασφαλούς ζώνης και μιας ασφαλούς περιοχής για τον χώρο ο οποίος είναι υπό τον έλεγχο των ε, αντιστασιαστών των επαναστατών κατά του Καντάφη είναι κάτι το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί διότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η ασφαλής ζώνη δεν βοήθησε αυτούς που βρισκόντουσαν εκεί αλλά αυτό ήταν το λάθος το οποίο διέπραξαν οι δυτικές χώρες. Άρα αυτή είναι η ιδέα την οποία αξίζει να εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες και ίσως αυτό θα επιτευχθεί στα πλαίσια του CACB. Επίσης, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε χώρες οι οποίες σήμερα δεν έχουν αναφερθεί δηλαδή δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τι γίνεται στο Μπαχρέιν σήμερα και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 Βέβαια ε, χαιρετίζουμε τις ε, ε, διαδηλώσεις που έγιναν στη Λιβύη και όταν εξετάζουμε τα οικονομικά βάδη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα για το κακό που έχει γίνει σε αυτές τις περιοχές. Ο κύριος Στάνο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ για την πρώτη δήλωσή σας από την Επιτροπή που αφορά σε αυτό το πολύ μεγαλεπίβολο σχέδιο βοήθεια Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Μεσόγειο. Η δική μου η ομάδα στηρίζει την ε, πολυμερή δημοκρατία στη Βόρεια Αφρική και τον Αραβικό κόσμο. Βεβαίω, η δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο αδιάβλητες εκλογές και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι η ε, Επιτροπή Εκλογών στην Τινησία αρνήθηκε να καταγράψει δύο Ισλαμικά κόμματα με τη δικαιολογία ότι ήταν ε, αντισυνταγματικά γιατί είχαν στην, στο προεκλογικό του ε, πρόγραμμα ε, διακριτική μεταχείριση ομοφιλοφίλων ε, γυναικών. Δεν πρέπει λοιπόν να ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ, και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να έχουμε τόσο ακραία κόμματα τα οποία δημιουργούν μια δημοκρατική πρόφαση. Ένα, εγώ είχα πει ότι πρέπει να υπάρχει ένα mini Marshall Plan για την Τινησία και τον επενδύσουμε εκεί. Αυτό αξίζει τον κόπο. Παρότι βέβαια αυτό ε, είναι αμφισβητούμενο από τους εκλογείς ε, ίσως ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μεταφερθούν κονδύλια από άλλες περιοχές από την ανατολική εταιρική σχέση αν συνέβαινε κάτι τέτοιο αυτό θα συνέμενε ότι θα υπήρχαν πάρα πολλοί οικονομικοί μετανάστες στην Τινησία έχει πάυσει τελείως ο τουρισμός οι ξένες επενδύσεις και αυτές κατόπιν τούτου στην περίπτωση αυτή θα προκαλούσαμε μια οικονομική κρίση που δεν νομίζω ότι θα τους βοηθούσε πρόθεσμα, ούτε και βραχυπρόθεσμα σε αυτή την προσπάθεια της ε, <clears throat> μετάβασης. Για τη Λιβύη ανησυχώ ιδιαίτερα ο Καντάφη και η ψυχοπαθήση, η γη του αν αυτοί επικρατήσουν αυτό θα προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση στη Λιβύη και επίσης και ένα εφιάλτη όσον αφορά την ασφάλεια στη Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θέλω να ελπίζω ότι όλα τα παγωμένα κεφάλαια οι λογαριασμοί του που έχουν παγώσει θα παραμείνουν παγωμένοι γιατί αλλιώς οι άνθρωποι θα πούν γιατί η Δύση και το ΝΑΤΟ θέλησε να σώσει τους Κούρδους και τους Κωσοβάρους, όχι όμως τους Λίβιους, οι οποίοι είχαν επίσης να αντιμετωπίσουν ένα τύρανο όπως είναι ο Καντάφη. Ο κύριος Φλότρε, ε, ε κυρία με συγχωρείτε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Εγώ διάβασα με μεγάλη χαρά την ανακοίνωση, αλλά αυτό ήταν πριν την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταλείψει στις ορδές του Καντάφη τους δημοκράτες της Λιβύης. Και σήμερα πραγματικά ε, ε, σπαράζει η ψυχή μας, διότι υπάρχουν ε, εκκλήσεις για βοήθεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να βοηθήσει τους δημοκράτες. Και είναι δύσκολο να λέμε αυτά τα οποία λέμε. Και αναρωτιέμαι εάν αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης των φοβερών επιπτώσεων που θα έχει αυτή η εγκατάλειψη στις βόμβες των Λιβύων επαναστατών και πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού οι οποίες διεξάγονται. Είναι τρομακτική κατάσταση Υπάρχουν 8.000 άτομα τα οποία θεωρούνται πρόσφυγες για το γραφείο της Τρίπολης. Ε, δεν συμμετέχουν στα προγράμματα διότι πολλοί έχουν φύγει αλλά δεν μπορούν να επανέλθουν στη χώρα τους και το πιο λογικό για τα άτομα αυτά είναι να βρούμε χώρες όπου θα μπορούν να εγκατασταθούν και πάλι. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί ε, να διαφημίζει την ε, επανεγκατάσταση αν η ίδια δεν πράττει αυτά τα οποία πρεσβεύει. Και νομίζω ότι είναι πολύ βλαβερό για την ε, συνεργασία την οποία εμείς θέλουμε να προωθήσουμε με, για, υπέρ της δημοκρατίας με τις χώρες της Νοτιού Όχθης της Μεσογείου. Ευχαριστώ κύριος Χουντής για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φούλε, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν με πείσατε ότι με τις μέχρι τώρα πράξεις και ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πράγματι βρισκόμαστε σε ένα ποιοτικό άλμα όπως ισχυριστήκατε σε σχέση με την αλλαγή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχέσεων με τις χώρες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση εξέγερσης και γενικότερα με τις χώρες της Μεσογείου. Και δεν με πείσατε γιατί Νομίζω ότι με αυτά που γίνεται, με τις θέσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διάβασα, ελπίζω αρκετά συστηματικά και τις 25 δράσεις που συζητήσατε νομίζω στην Κομισιόν και που αφορούν όλες αυτές τις χώρες. Η γεύση που μου δώσατε είναι όπως κατά το πρόσφατο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαζόταν με αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα, τα στήριζε, έχει ευθύνη για τη μακροημέρευσή τους, έχει ευθύνη για την κατάσταση που έφτασαν προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, σήμερα γίνεται μια απόπειρα να ηγεμονεύσει ή να κυριαρχεί στις εξελίξεις, ορισμένες μάλιστα είναι σαν να τις υπαγορεύουμε κατά τις δικές μας απαιτήσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα ίδια συμφέροντα. Φοβάμαι πως είμαστε στην ίδια κατεύθυνση κύριε Φούλα και γι' αυτό νομίζω ότι δεν έχω πιστεί νομίζω ότι πράγματι δεν έχει αναθεωρηθεί η κακή, λαθεμένη, αποτυχημένη πολιτική γειτονία που ακολουθήθηκε σε αυτή την περιοχή. Θέλω να σας πω ε, επιπρόσθετα και επικουρικά. Εδώ υποτιμάται το γεγονός ότι αυτοί οι εξεγέρσεις δεν είναι μόνο απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα που είναι και που πρέπει να τα καταδικάσουμε και που είμαστε αντίθετοι έχουν και οικονομικές και κοινωνικές διεκδικήσεις. αυτοί οι λαοί ζητάνε καλύτερο μέλλον καλύτερο οικονομικό και κοινωνικό μέλλον και η δική μας μέχρι τα τώρα πολιτική αλλά και ο σχεδιασμός μάλλον δεν προϊονίζεται ότι πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, δεν φαίνεται με υποκριτικές τάσεις να αναλαμβάνονται ευθύνε για το πρόβλημα της μακροημέρευσης και της αμφίδρομης διαφθοράς που υπήρχε μεταξύ αυτών των κατεστώτων και πολιτικών ηγεσιών στην Ευρώπη. Θυμίζω και τελείωσα τις σχέσεις που αποκαλύπτονται αυτή την περίοδο μεταξύ της ηγεσίας της Λιβύης και του Προέδρου Σαρκοζή οι καταγγελίες ότι ε, ο προεκλογικός αγώνας ενισχύθηκε από τους Λίβιους. Επομένως υπήρχε αμφίδρομη διαφθορά, πράγμα που πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά. E Μίλησαν λοιπόν οι πολιτικές ομάδες ε, και θα έχουμε τώρα για ένα λεπτό μόνο οι επόμενοι ρωτώντε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να ε, σας αναφέρω μια δική μου παρατήρηση, λέει ο κύριος Πρέντα. Ε, συμφωνούμε όλοι ότι ε, στον τομέα της δημοκρατίας, της οικονομίας και της στήριξης των πολιτών είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία. Αλλά όπως υπογράμμισαν και οι συνάδελφοί μου, εκτός από αυτή τη συμφωνία θα πρέπει να ορίζουμε καλύτερα τα κριτήρια. Έχω λοιπόν να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά στο θέμα της διαφοροποιημένης προσέγγισης των κρατών. Ε, θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον προτίθεστε στο εγγύς μέλλον να εγκρίνετε ένα πρόγραμμα που να αφορά σε μια καλύτερη γειτονία, πολιτική γειτονία με αυτές τις χώρες το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάει για λάθη, όμως δεν αναφέρεται καμία λύση, έτσι ώστε να έχουμε μια ε, καλύτερη στάση ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στη Μεσόγειο. Ευχαριστούμε. Κυρία Γκόμες, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η ανακοίνωση είναι πολύ καλή, κύριε Επιτρόπε. Αλλά δεν θα αξίζει το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένοι, αν αποτύχουμε στη Λιβύη. Θα πρέπει να πείτε την κυρία Άστον ότι αν δεν κάνουμε τίποτα στη Λιβύη και αν δεν αποτρέψουμε το καθεστώς του κατάφη να ε, κατασφαγιάσει τον κόσμο στη Βεγγάζη, καλύτερα να μείνει και που είναι η κυρία Άστον. Αναφερθήκατε στις επιχειρήσεις, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που από ό,τι φαίνεται φοβούνται ότι θα επηρεαστούν από το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων. Μα η κοινή γνώμη υποψιάζεται ότι γι' αυτό ακριβώ το λόγο καθυστερούμε και κολυσιεργούμε και δεν αναλαμβάνουμε δράση στην ε, ε Λιβύη γιατί σιωπούμε μπροστά στην εισβολή της Σαουδικής Αραβίας στο Μπαχρέιν. Γιατί δεν είχαν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του Μομπάρακ. Θα πάμε, θα στείλουμε κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο. Θέλουμε απάντηση γι' αυτό. Θα ήθελα να πω εκ μέρους της κυρίας Φλότρου να Βατάνεν που όλα αυτά τα χρόνια είχαν α, ε, σχέσεις ε, με αυτούς τους γενναίους ανθρώπους που δίνουν μάχη υπέρ της δημοκρατίας στην περιοχή αυτή του κόσμου. Το Κοινοβούλιο νομίζω ότι μπορεί να στηρίξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αφήσει το λαό στη μοίρα του. Ο κύριος Μιγιάν Μόν για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι για το νέο προσανατολισμό που θα δώσετε στην πολιτική γειτονία και θα διαβάσω με ιδιαίτερη προσοχή την νέα ανακοίνωση, γιατί τη φιλομέτρησα προς το παρόν ακροθυγός. Δυναμική είναι η προοπτική, υποστηρίζει τις ε, εξελίξεις ή τις επαναστάσεις ε, που θα οδηγήσουν σε πραγματικά δημοκρατικά καθεστώτα και ελπίζω για να δοθεί το αναβαθμισμένο καθεστώς να συντρέχουν μια σειρά προϋποθέσεων. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο. Το εμπόριο σίγουρα είναι ένας τρόπος δημιουργίας πλούτου και στις διόχθες της Μεσογείου. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι σημαντικό και το θέμα των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες αυτές, τις χρηματοπιστωτικές ροές. Και ως προς το εμπόριο, ρίξτε μια ματιά στην έκθεση που υιοθετήσαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και έχει τίτλο «Γεωργία και Διεθνές Εμπόριο». Γιατί πολλοί γεωργικοί τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι αυτοί πληρώνουν τα σπασμένα και είναι το θύμα στο βωμό της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και αυτοί είναι που χάνουν τις συμφωνίες. Γιατί μιλούμε για, για κοινωνικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές προδιαγραφές θα πρέπει να πληρούνται πριν καταλήξουμε στη σύναψη των συμφωνιών. Και πραγματικά δεν θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η διακριτική μεταχείριση βάρο των γεωργών του αγροτικού κλάδου και υπέρ ορισμένων άλλων κλάδων. Κύριο Κυρίλοφ, για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε. Πολύ σύντομα. Ε, θέλω να πω ότι σας στηρίζω ανεπιφύλακτα σε όλα αυτά που προτείνετε. Απλά θα ήθελα να τοποθετηθώ, ε, μάλλον όπως και η συναδελφοί μου και εγώ να σας ζητήσω να αντιδράσετε σε ένα πιθανό ρεαλιστικό σενάριο. Μετά από λίγες μέρες ας υποθέσουμε ότι οι δυνάμεις ε, του ε, Καντάφη φτάνουν στη Βενγάζη, στο προπύργιο των, ε, των εξεγερθέντων και θα έχουμε αναμφίβολα αιματοχυσία. Έχουμε λοιπόν τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά σκάφη μπροστά από τη Βεγγάζη σε διεθνή ύδατα. Ως πολιτική λοιπόν τι θα του πούμε. Έχουμε δύο δυνατότητες. Η μία εξ αυτών είναι να εμπλακούμε και να προσπαθήσουμε να σώσουμε από τους ανθρώπους ανεξάρτητα με το αν θα υπάρχει απαγόρευση υπερπτήσεων ή όχι. Η άλλη λύση αν πούμε γρήγορα, φύγετε γρήγορα. Γιατί ε, το να ε, βλέπει κανείς ότι διαδραματίζεται και το τι θα διαδραματιστεί θα είναι κάτι το ε, τρομακτικό, το παράδεκτο. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυρίλοφ, ε, Ουγγουριάνο, ε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, κύριε Επίτροπε, στις 16 Φεβρουαρίου η Ισπανία και μετά η Ισπανία, η Κύπρος και η Μάλτα απευθύνθηκαν στη Lady Άστον και είπαν ότι ο Νότος δεν, έχει, δεν λαμβάνει αρκετά κονδύλια και δεν θα πρέπει να αντιστραφεί η σχέση εις βάρος της Ανατολής. Αυτό όμως είναι λάθος ο ισχυρισμό, γιατί τα στατιστικά δεδομένα είναι λάθος, στέλνει ένα καταστροφικό μήνυμα ε, προς Ανατολάς και δημιουργεί και έναν ε, στρεβλό ανταγωνισμό ανάμεσα ε, στην Ανατολική και την νότια πλευρά της Ευρώπης. Εσείς λοιπόν τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε για αυτό το θέμα και στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας. Ευχαριστούμε και την συζήτηση θα ολοκληρώσει με ερώτηση η κυρία Λοκ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, εμείς ε, τα βασικά στοιχεία της ε, έκθεσής σας ε, που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα συζητήσαμε και δεν βρήκαμε απαντήσεις. Το ένα είναι αυτό που είπε η κυρία Φλότρε. Δηλαδή τι θα γίνει με τους μετανάστες από τη Σομαλία και την Ερυθρέα όπου η Επιτροπή Προσφύγων το ΟΗΕ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιληφθεί του θέματος και να βοηθήσει να απομακρυνθούν από τις ε, γενέτηρές τους, από τις αιστείες τους. Η Frontex έχει ως καθήκον να προστατεύεται στην ώρα αλλά και να βοηθάει. Πώς αυτά συμβαζίνονται με τη την ε, δήλωση, με την πληροφορία που υπάρχει σήμερα στο Financial Times όπου η Ιταλία αρνήθηκε να ε, δεχθεί ένα πλοίο που ερχόταν από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Εσείς λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε οι πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές να γίνονται αποδεκτοί στη δική μας την περιοχή. Εντάξει λέει ο πρόεδρος, ε, έχουμε ακόμα τέσσερα λεπτά πριν από ε, την ε, εκπνοή του χρόνου μας. Και έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης που με ακούσατε στην αρχή και ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι σωστό είναι να λεχθεί και να επαναληφθεί ότι αυτά τα οποία διαπιστώνουμε εις τη νότια όχθη της Μεσογείου είναι τρομακτικά και βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις πρωτεύουσες των κρατών μελών, στις Βρυξέλλες και στο Συμβούλιο των Υπουργών και στο Κοινοβούλιο όντως ε, προκάλεσε και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να ε, χαρακτηρίζεται από τα ίδια στοιχεία και τις ίδιες αρχές. Προτού προχωρήσω σε συγκεκριμένα σχόλια είμαι βέβαιος ότι εσείς είστε καλύτερα, θα είστε, πιο κατάλληλοι να θέσετε αμε, αμέσως τα ερωτήματά σας στην κάθε άστον. Διότι εγώ, ε, ναι μεν συμφωνώ με πολλά από τα σχόλιά σας, αλλά υπό αυτά στα συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να σχολιάσω αυτά που είπατε. Να ξέρετε όμως ότι δεν φύγω και θα χρησιμοποιήσω κάθε ευκαιρία η οποία μπορεί να μου δοθεί ε, σε περιορισμένο κύκλο χωρίς να εκφράζω πολιτική προτίμηση να συζητήσω εκτενώς τα θέματα αυτά. Η έκθεση την οποία παρουσιάζω σήμερα προσβλέπει προς το μέλλον. Μ' αρέσει να κοιτώ προς το μέλλον και έκανα σήμερα ορισμένα σχόλια και ε, άλλα σχόλια προηγουμένως για τους τρόπους με τους οποίους νομίζω που μπορούν να υπάρξουν συμβιβασμοί για να βελτιωθεί η αντιμετώπιση μας. Αλλά με τη βοήθειά σας και εδώ όντως θέλω να προσφέρω μία συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικοδομητική πρόοδο να συνεργαστούμε διότι πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχουμε απαντήσει μόνο στα εύκολα ερωτήματα. Έχουμε απαντήσει μόνο στο τι είναι έτοιμη να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε περίπτωση νοτίων γειτόνων σε χώρες οι οποίες ήδη ξεκινούν μία διαδικασία εκδημοκρατισμού. Ενώ υπάρχουν άλλα πιο δύσκολα θέματα. Τι θα γίνει με τις χώρες οι οποίες μόνο μονοπροσποιούνται ότι θα τροποποιήσουν την κατάσταση. Τι θα γίνει με τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή και είναι βασικό να καταλάβουμε όλοι ότι η ανακοίνωση που προσπαθούμε να υιοθετήσουμε σήμερα δεν γίνεται αποδεκτή με μονομένα. είναι μέρος της ευρωπαϊκής αναθεωρητικής διαδικασίας γυτνιάσεως και ε, της απάντησης σε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε επίσης να απαντήσουμε στις ερωτήσεις τις οποίες ήδη έφυξα σε αυτή την Επιτροπή και πέραν της μίας φορά. Δηλαδή ποιο, ε, το τελικό κέρδος της συνεργασίας μεταξύ ε, Ανατολών και Νότου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι αυτό το μέσο και συγχρόνως ε, σε συνδυασμό με, μια στρατηγική, με ένα στρατηγικό όραμα. Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Εγώ από τη μία πλευρά δεσμεύομαι προς το Κοινοβούλιο και προς την Επιτροπή σας. Ε, επίσης πέραν αυτού Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να ε, εφαρμόσει μια πολιτική γυτνιάσεως. Αυτό έχει λεχθεί και από τον πρόεδρο Μπαρόζο ότι θα υπάρξει και μια δεύτερη μονάδα που θα καθοριστεί από την πολιτική γυτνιάσεως και χαίρομαι διότι βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διότι δεν είμαι μόνος αρμόδιος αλλά βλέπω ότι όλο και περισσότεροι συνάδελφοι στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και τέλος, ε, στην διατύπωση κάποιου μέσου θα μπορέσουμε ε, να χρησιμοποιήσουμε επικοδομητικά τα, τους σπόρους μας, τους σπόρους μας προς συμφέρον μας. Όχι άτακτα προς τη μία κατεύθυνση από εδώ και την άλλη από εκεί αλλά θα ε, ζητήσουμε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως, την ΤΕΦΚΟ και άλλες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν καθημερινή διαβούλευση κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι αξίες μας και τα συμφέροντά μας θα καλύπτονται από αυτή τη νέα πολιτική Σήμερα ζήτησα από το συλλογικό όργανο, από τον πρόεδρο και από τους συναδέλφους να παρακολουθήσουν την εφαρμογή αυτής της ανακοινώσεως που παρουσιάσαμε στις 8 Μαρτίου διότι έχουμε εντοπίσει τα βασικά μέτρα είπαμε ποιος θα είναι υπεύθυνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τηλεγραφικά είπαμε και πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Ζητήσαμε επίσης από το συλλογικό όργανο να ε, διατυπώσει μία δικούσα επιτροπή η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται συντονισμένα και εκεί θα εκπροσωπείται και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, σήμερα ξεκινήσαμε μία σημαντική και αναγκαία διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή προσπαθούμε να εξετάσουμε τα εθνικά προγράμματα ενδεικτικά από όλους τους γείτονές μας ιδίως στο Νότο και Ανατολάς και ε, να δούμε πού βρισκόμαστε δηλαδή να δούμε πού θέλουμε να ενταχτούμε και αν δούμε ότι το πρόγραμμα δεν συνάδει με αυτά τα οποία εμείς επιθυμούμε ε, θα ε, ε, εστιαστούμε στα θέματα αυτά θα επανέλθω σε αυτό το, εδώ στο Κοινοβούλιο και θα συμμετάσχω στα πλαίσια κάποιες εκδηλώσεις που εσείς θα επιλέξετε στη συζήτηση των θεμάτων αυτών μαζί σας κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορείτε να είστε βέβαιοι και να γνωρίζετε ότι με πλήρη διαφάνεια κάνουμε αυτά τα οποία δεσμευόμαστε να κάνουμε και διακηρύσουμε ότι θα κάνουμε. Όσον αφορά ορισμένα ερωτήματα του κυρίου Σαλαφράγκα για την αναθεώρηση της χρηματοδότησης, πέραν της κινητοποιήσεως των πόρων για να καλύψουμε τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, εξετάζουμε τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα και εδώ δεν μιλάμε για πενταροδεκάρες, μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2011 ως το 2013 για όλη την περιοχή. Επίσης εξετάζουμε την, τις επικεφαλίδες των τομέων. Δεν είναι χρήματα τα οποία είναι στην πάντα και περιμένουν πώς θα εφαρμοστούν, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τα διάφορα προγράμματά μας, να τα συγκρίνουμε τις ανάγκες των συναδέλφων μας και γειτόνων μας και να δούμε ε, χρειαζόμαστε τους πόρους αυτούς, ε, μπορούμε να τους αφήσουμε αδρα αυτή τη στιγμή ή θα τους χρησιμοποιήσουμε καλύτερα εάν τους χρησιμοποιήσουμε για την πολιτική γενιάσεω. είναι ίσως πολύ, πολύ νωρίς για να αποφανθούμε αλλά ένα μέρος από αυτά τα χρήματα αντιπροσωπεύει σημαντικούς πόρους και επιπλέον Ε, πρέπει να βρεθούν οι πηγές χρηματοδοτήσεως και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πώς ε, ε, θα κινηθούμε καινοτόμα για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την, τις δυνατότητες επενδύσεως διότι μόλις η διαδικασία αυτή ξεκινήσει Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να έρθω σε επαφή μαζί σας και να σας ενημερώσω για το ύψος των κεφαλαίων τα οποία θα χρειαστούν. Ε, η κυρία Ντεκάιζερ είχε μία πολύ ε, σημαντική ερώτηση για το μηχανισμό. Σας είπα ότι ελπίζω ότι ως την επόμενη συνάντησή μας θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω ότι λειτουργεί σωστά. Δεν θα ρωτήσω μόνο ο, τους γραφειοκράτες των Βρυξελών αλλά και τα ελπίζω ότι οι ριζικές αλλαγές τις οποίες διαπιστώνουμε με την ε, ρεαλιστική πολιτική ε, θα οδηγήσει στις ε, σωστές πράξεις που θα ακολουθήσουν τις σωστές διακηρύσεις διότι έχουμε τον μηχανισμό ξέρουμε πως μπορούμε να τα κάνουμε σωστά τα πράγματα αλλά ε, και όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικά θέματα. Κύριε Πρόεδρε, Ετέθη επίσης ένα ερώτημα μεταξύ άλλων ε, για την ομάδα των ε, προσφύγων, για τους πρόσφυγες και για όλους εκείνους που έχουν χαίρουν ειδικού καθεστώτος. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Παρασκευή παρουσίασα το θέμα και την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα αυτό ετέθη στο κολέγιο των επιτρόπων και στους αρμόδιους επιτρόπους η αρμόδια επίτροπος δεσμεύτηκε να έρθει σε επαφή με τα άμεσα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη και να βρει μια λύση για όσο δυνατόν περισσότερους πρόσφυγες. Από όλα αυτά λοιπόν που σας είπα φαντάζομαι ε, θα μπορούσατε να συνάγετε ότι αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν τάσσομαι υπέρ του να μετακινηθούν οι πόροι από ε, την ανατολική πλευρά της Ευρώπης προς τον Νότο. Φαντάζομαι όμως ότι θα έχετε κατανοήσει ότι είμαι υπέρ του να ε, μεταφέρουμε κονδύλια εκεί που υπάρχει δράση και δράση ενώ υπάρχει διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Έχουμε δύο ε, διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης και όπως και οι υπόλοιπη Ευρώπη ε, σκέπτονται τις αλλαγές στον Νότο, έτσι θέλω να πιστεύω και οι ανατολικές περιοχές θα προβληματιστούν και αυτές και θα προβούν σε βέλτιστη χρήση των πόρων των οποίων, ε, τους οποίους ε, λαμβάνουν. Όσον αφορά τώρα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αυτό είναι μία από τις τελευταίες ερωτήσεις που ετέθησαν. Ε, είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εγώ έχω ήδη αφήσει να εννοηθεί στους συναδέλφους μου ότι είμαι πρόθυμος να ε, απευθυνθώ ε, στην Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να προβάλλουμε το πόσο σημαντικό σημαντικά είναι αυτά τα θέματα έτσι ώστε και η πολιτική μας να είναι και πιο σωστή. Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να κλείσω με αυτά τα λόγια. Πάρα πολύ καλά, λέει ο Πρόεδρος όχι ήσασταν, δεν ήταν μόνο ακριβής αλλά και πολύ περιεκτικός και τουλάχιστον όσον αφορά εμάς ε, θεωρώ ότι είσαστε ένας από τους επιτρόπους ε, εκείνους ε, που είναι, επιδεικνύουν ιδιαίτερο πνεύμα συνεργασία με την Επιτροπή μας ε, και βεβαίως ε, πράγματι εξαντλήσατε τα θέματα αυτά που ετέθησαν περίπλοκα πολύ θετική η σημερινή μας συνάντηση όπως και όλες οι άλλες που έχουν προηγηθεί και είμαι σίγουρης και εκείνες που θα ακολουθήσουν ε, ας ευχηθούμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο θα συνεχιστεί η σχέση μας και θέλω να πιστεύω ότι και εσείς ακούσατε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, ε, κάποιες απόψεις ε, για να ε, συνεχίστε να αναλαμβάνετε, να εξασκείτε, να ασκείτε με συγχωρείτε, με υπευθυνότητα τα καθήκοντά σας. θα ξανασεντούμε στις 22 Μαρτίου στις 9 ώρα το πρωί, λίγη στην συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ.